Okay, those colleagues who here, just to make the point the start. Καλή σας μέρα. Είναι τρεις αγαπητοί συνάδελφοι και επομένως θα ε, ξεκινάσω. Θα ξεκινήσω και αυτοί οι οποίοι θα έρθουν ας έρθουν με την ησυχία τους. Τι θα τους κάνω εγώ. Σχέδιο ημερήσιας διάταξης λοιπόν το εγκρίνουμε. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω ε, αυτήν την ομάδα από την Τυφλίδα την, ε, ε, της γεωργίας είναι φοιτητές, του έφερε ο κύριο Σέτσο. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι στην τελευταία Eurovision εγώ ψήφισα το, το τραγούδι της Γεωργίας. Uh, λοιπόν, όταν θα πάτε στην ε, Γεωργία, θα πείτε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών θεώρησε ότι το καλύτερο τραγούδι στην Eurovision ήταν ε, οπωσδήποτε αυτό της Γεωργίας. Θαύμα. Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, επαλήθευση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος από τις θαλάσσιες μεταφορές και τροποποίηση κανονισμού Μίκαελ Κράμερ. Έχεις το λόγο. <laughs> Λοιπόν, οι πλωτές μεταφορές είναι ο μόνος τομέας, ή συγχωρείτε, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο μόνος τομέα που δεν έχουν οι εκπομπές ρήπων συμπεριληφθεί και αυξάνονται και αν δεν αλλάξει τίποτα το, το, το 2020 θα έχουμε μια τεράστια αύξηση και αυτό όχι μόνο βλάπτει το κλίμα αλλά και την υγεία διότι έχουμε και 50.000 πρώιμους θανάτους που οφείλονται στην ρήπανση της ατμόσφαιρας από τις ναυτικές ναυτιδιακές μεταφορές. Λέει πολλά πράγματα η IMO, αλλά δεν κάνει αρκετά. Υπάρχουν επίσημοι δείκτες, αλλά δεν είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Για κάποιες νέες κατηγορίες πλοίων και για κάποια σχέδια διαχείρισης των στόλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν όπως έχουν προβλεφθεί και πρέπει να επιτευχθεί 40% ή και 50% των εκπομπών ρήπων σε σχέση με το 2005. Ήταν η έκθεση Gross, θέλω να το υπενθυμίσω. Είχαμε συζητήσει διεξοδικά και για τις επιμέρους κατηγορίες υπήρχαν πολλοί προσανατολισμοί, κατευθυντήριες γραμμές. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. Τώρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να ακολουθήσει η δράση. Και τώρα δεν σέβεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στη ρύθμιση ενός τέτοιου συστήματος μέχρι το 2030, να το επεκτείνει και αν μέχρι το 2011 δεν θα έχει υπάρξει μια διεθνή συμφωνία, ήταν μεγάλες οι φιλοδοξίες. Αλλά για τις εκπομπέ ρήπων στι εναέριες μεταφορέ υπήρξε τέτοια, ας το πούμε έτσι, ε, τέτοιο θάμβος που δεν ε, μπόρεσαν να γίνουν άλλα πράγματα. Η γνωμοδότηση και οι διαπραγματεύσεις. Ήταν δυσχερείς οι διαπραγματεύσεις διότι οι θέσεις μας ε, παρεξέκλειναν πολύ και ήταν τόσο μεγάλες οι διαφορές, σημαντικό είναι και πρέπει να το πούμε ότι πρέπει να το εγκρίνουμε αυτό, αυτό το οποίο και το, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε η συνεπής ε, ένταξη των πλοίων σε σχέση με την ε, χωρητικότητά τους, ε, κόρων ολικής χωρητικότητας, gross και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και οι άλλες βλαπτικές ουσίες να συμπεριληφθούν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις εκπομπές θείου Αυτά τα δύο σημεία πολύ σημαντικά και παρακαλώ λοιπόν ως εισηγητής και πάλι να εγκρίνετε να τα καταφέρουμε να προχωρήσουν αυτά, να μην μείνουμε πίσω από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο εισηγητής, ε, ο κύριος Σκυλακάκης ε, από την Ελλάδα, φιλελεύθερος, υποστηρίζει αυτή τη θέση. Ήταν κάπως εκπληκτικό για αρκετούς από εμά και το λέω και το τονίζω και μετά από ερώτηση που του έγινε είπε ότι πράγματι δεσμεύεται Τώρα, φαντάζεται κανείς ότι είναι μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τις ε, εκπομπές ρήπων στις ε, εναέριες μεταφορές ε, ο μεγαλύτερος αντίπαλος ήταν η ΕΠΑ και σε σχέση με την ε, ένταξη αυτών των ε, πλοίων όσον αφορά ένα ε, πλαίσιο το οποίο δεν θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε χειρότεροι από τις ΣΥΠΑ πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν να μην ξεχνάμε την οικονομική, το οικονομικό κέρδος το οποίο είναι μεγάλο δεν πρόκειται μόνο για την οικολογία αλλά και για την οικονομία που είναι σημαντικό αυτό το θέμα και περιγράφεται και αντίστοιχα και αν με την υφιστάμενη τεχνολογία για, ε, για τα μέτρα αυτά οι εκπομπές ε, ρήπων ε, διοξιδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 75% και με μείωση της ταχύτητας 10% στην μεταφορά αγαθών δεν παίζει ρόλο η ταχύτητα αλλά παίζει ρόλο ο χρόνος παράδοσης. Πρέπει να δούμε αν κάποιος βρίσκεται 20-24 ώρες καθοδόν αυτό δεν παίζει ρόλο πρέπει η ώρα να είναι σωστή στην παραλαβή και παράδοση. Ωστόσο όμως ε, σε σχέση με τις, ε, με μεταφορές με τα πλοία πρέπει να δούμε τα κόστη τα οποία είναι υψηλά με υψηλές ταχύτητες και πρέπει να δούμε όχι μόνο το, την αυτή οικονομικά αλλά και σε σχέση και με το περιβάλλον. Συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτά τα σημαντικά συμπεράσματα. Η ναυτιλία πρέπει να συνεισφέρει ώστε μεταξύ των άλλων ε, φορέων μεταφορών να ενταθούν και οι θαλάσσιες μεταφορές. Ένα σαφές μήνυμα να δοθεί ότι σε αυτά τα σημεία υποστηρίζουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και έτσι ευχαριστώ και για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στους ε, ε, σκιώδεις, τον κύριο Σερβάν από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Τι να πω. Το ΕΛΚΑ... πρώτα απ' όλα ευθυγραμμίζεται με την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κατά την άποψή μου πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα και σφαιρικά. Αυτό στη δικιά μου γλώσσα και το δικό μου μυαλό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι μπορούμε να επιτύχουμε βάζοντας αυτά τα όρια για τους 400 τόνους. Ε, περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερο γραφειοκρατικό κόστος. Ε, τι θα επιτύχουμε όμως ε, και όσον αφορά το περιβαλλοντικό όφελος και ποια θα είναι τα απτά αποτελέσματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσουμε και τη θέση των ναυτιλιακών εταιριών και επομένως πιστεύουμε ότι η πρόταση της ε, ε, Κομισιόν είναι μετριοπαθής, όντως. Δεν είναι πολύ φιλόδοξη. Αλλά είναι και ρεαλιστική πρέπει να πω. Έχουν κάποιους λόγους που κρατάνε αυτό το βάρος τους 400 τόνους. Ε, είναι τα 55% των πρωτοκόλων που σημαίνει ότι αυτά τα πλοία αντιπροσωπεύουν περίπου 90% του συνόλου. Υπάρχει λόγος λοιπόν που κρατάει το ε, κατόφλι του βάρους ε, εκεί. Γιατί από εκεί και πέρα θα μπορούσε να βαρύνει πολύ την γραφειοκρατία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές θα πρέπει να δούμε επίσης ότι η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από την IMO. Και το πεδίο εφαρμογής, τελευταίο αλλά σημαντικό, πιστεύουμε ακριβώς ότι επειδή η, το, διοξίδιο του, το διοξίδιο του άνθρακα αντιπροσωπεύει το 9, τα 9 δέκατα της ε, μολύνσης, θα πρέπει να τα κρατήσουμε τα επίπεδα εκεί δεν ξέρω αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, συνένεση για τους 400 τόνους, αλλά ε, σίγουρα δεν μπορούμε να φτάσουμε στις 5.000 ε, τόνους. Αλλά 500 τόνους μπορούμε να φτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάκενστάιν από τους Σοσιαλιστές. Πρόεδρε, και εμείς ευχαριστούμε τον εισηγητή, το συντάκτη γνωμοδότησης για τη μεγάλη προσπάθειά του, ακόμα και αν διαφωνούμε με κάποια σημεία μαζί του. Είναι σημαντικό η ναυτιλία και αυτή να συνεισφέρει. Είναι επίσης σημαντικό από τον τομέα των εναέριων, μεταφορών να συναγάγουμε μαθήματα και να μην επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα στην ναυτιλία μια και η εποπτεία θα βρίσκεται εκτός των ε, ε, υδάτων της επικράτειας των κρατών μελών σε σχέση με τα πλοία και σημαίες τρίτων χωρών θα πρέπει να διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι τρίτες χώρες δεν θα υποβάλουν θέματα επιφύλαξης ε, και θα μπορέσουμε έτσι να καταβάλουμε προσπάθειες να γίνει διεθνώς αποδεκτό αυτό το εγχείρημα. Είναι σημαντικό ένα καλό βήμα αυτό από ευρωπαϊκής πλευράς ώστε παγκόσμια να προαχθεί αυτό το θέμα και να έχουμε και ένα μηχανισμό μηχανισμό που θα βασίζεται στην αγορά για αυτές τις ε, εκπομπές. Αν θέλουμε να έχουμε μια παγκόσμια τέτοια συμφωνία, σφαιρική συμφωνία, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συμβατότητα την συμβατότητα του κανονισμού με διεθνείς άλλες συμφωνίες να την εγγυάται και να την διασφαλίζει. Συγκεκριμένα τώρα για τα πεδία εφαρμογής όσον αφορά το μέγεθος των πλοίων συμφωνούμε με τον εισηγητή στην πρότασή του και θα είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε το συμβιβασμό συνολικά δηλαδή να δεχθούμε το συμβιβασμό και μικρότερα πλοία από 400 τόνους να συμπεριλαμβάνονται. Όσον αφορά τα πεδία εφαρμογής, όσον αφορά τις βλαπτικές ουσίες Μέχρι σήμερα προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιορίζεται στο διοξίδιο του άνθρακα η πρόταση και συμφωνούμε με αυτό το πλαίσιο. Μέχρι τώρα και μέχρι τη σημερινή χρονική στιγμή. Θα ζητήσουμε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διετή περίοδο να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση για τις τεχνικές προόδους, την τεχνική πρόοδο και δυνατότητα να ενταχθούν και άλλες βλαπτικές ουσίες σε αυτή την πρόταση. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι 98 περίπου είναι 98% όλων των αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με την, ε, τις θαλάσσιες μεταφορές. Και μια μελέτη του IMO λέει ότι το διοξίδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο αέριο όσον αφορά την ε, ναυτιλία και σε σχέση με την εκπομπή ρήπων σε άλλα αέρια είναι περιορισμένη καθώς επίσης και όσον αφορά τον όγκο και όσον αφορά και το, ε, την δυνατότητά τους να επιτυγχάνεται ε, θέρμανση, υπερθέρμανση του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει λοιπόν ότι άλλου είδους τέτοια αέρια δεν θα συμπεριλαμβάνονται και θα πρέπει να ενταχθούν με τρεις ε, μονάδες συσκευές μέτρησης που είτε μέχρι σήμερα δεν ήταν αξιόπιστες είτε ήταν υπερβολικά δαπανηρές και όλα αυτά δεν φαινόταν να είναι αποτελεσματικά. Λοιπόν, αν συμβαίνουν όλα αυτά θέλουμε να ακούμε ένα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διετή περίοδο αν κάτι έχει αλλάξει, αν έχει σημειωθεί πρόοδος και αν έχει νόημα να συμπεριληφθούν και τα άλλα αέρια. Οι τέσσερις μέθοδοι για τη μέτρηση που προτείνονται πρέπει να τηρηθούν πιστεύουμε. Ωστόσο όμως σύμφωνα με την, με, σε τακτά διαστήματα θα πρέπει να μας υποβάλει συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας λέει αν είναι δυνατόν να μειωθούν αυτές οι εκπομπές περαιτέρω και θα πρέπει το δυνατόν γοργότερα να αρχίσει να ισχύει αυτή η ρύθμιση ώστε να υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθούμε και να συνεισφέρουμε στη μείωση εκπομπών ρήπων. Αυτά είναι συντομία η δική μας γνωμοδότηση, η δική μας τοποθέτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σαμισά για τους φιλελεύθερους. Έχουμε ένα πρόβλημα διερμηνίας. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μπορούμε... Μήπως θα μπορούσατε να αρχίσετε από την αρχή. λειτουργούν τώρα όλα. Εντάξει, επιλύθηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ τον συντάκτη γνωμοδότησης. Δεν είναι καθόλου απλό το ζήτημα αυτό και δεν υπάρχουν και απλές λύσεις ε, σε αυτά τα προβλήματα. Όσον αφορά την ουσία του θέματος, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν εκείνη που αναμέναμε και προσδοκούσαμε. Οι στόχοι δεν ήταν επαρκείς. Κυρίως επειδή εδώ πρόκειται μόνο για τις εκπομπές τρύπων διοξιδίου του άνθρακα μόνο και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για μείωση. Δεύτερον, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, διαρκεί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό. Και τρίτον, πρόκειται πάλι εδώ μόνο για διοξίδιο του άνθρακα λοιπόν σε αυτές τις εκπομπές ρήπων. Εδώ το τα οξύδια του αζότου και άλλες βλαπτικές ουσίες ε, δεν έχουν ενταχθεί, έχουν παραμεληθεί. Υποβάλλει λογικές προτάσεις ο συντάκτης γνωμοδότησης. Θα πρέπει να είναι όμως συντομότερο το χρονοδιάγραμμα και όλες οι εκπομπές ρήπων, όλα τα αέρια που ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα να συμπεριληφθούν και αυτά. Είναι σημαντικό και το θείο και τα οξύδια του θείου να ενταχθούν. Αυτό που θέλουμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες εξειδικευμένες προτάσεις ε, για την μείωσή τους. Πώς θα γίνει αυτό, αυτό θα το αποφασίσει και θα το κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό δεν μπορούμε σε σχέση με αυτό να υποστηρίξουμε τις ε, προτάσεις. Ε. Όσον αφορά την αυτιλία γενικότερα, υποστηρίζουμε τους στόχους του συντάκτη γνωμοδότησης και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι το 400 ως σημείο αναφοράς είναι σημαντικό στοιχείο, όπως προβλέπεται και από τον IMO, τον Διεθνή Οργάνωση Ναυτιλίας. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούμε λοιπόν για το ότι τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται και έτσι δεν, υπάρχει, δεν θα υπάρχει πρόσθετο κόστος για τους εφοπλιστές και πλειοκτήτες. Ευχαριστώ. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής μου ομάδας. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τους ε, Ευρωπαίους Μεταρρυθμιστές, ο κ. Βαντάλεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μας, Πρόεδρε, θα θέλαμε να παραμείνουμε κοντά στην ε, πρόταση της Επιτροπής Τη θεωρούμε εξαιρετική. Ο εισηγητής κινείται προς μια κατεύθυνση στην οποία δεν μπορούμε να στερήξουμε. Θεωρώ θετικό σημείο βέβαια ότι μιλά για την ποιότητα των καυσίμων, γιατί δάλλως πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα ε, με διάφορα μείγματα καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αυσεπλοεία. Σε αυτό λοιπόν το στερίζουμε, αλλά κατά τα λοιπά μας δημιουργεί πρόβλημα η γραμμή που ακολουθεί ο εισηγητής και θα προτιμούσαμε να παραμείνουμε όσο δυνατόν πιο κοντά στην πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Στρέφουμε τώρα προς την Επιτροπή. Κυρία Μπάτζαμ, από την Γενική Διεύθυνση Εκκληματική Αλλαγής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου που παρενέβησαν. Νομίζω ότι σιγά σιγά εντοπίζουμε τα στοιχεία της συζήτησης. Θα ήθελα λοιπόν ε, σε δύο λεπτά να σας ε, παρουσιάσω τη δική μας οπτική γωνία. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, πάντα θεωρούσαμε ότι το να επικεντρωθούμε στο διοξείδιο του άνθρακα ως ε, βασικό ρήπο είναι η κατάλληλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες ε, τεχνικές τουλάχιστον προκλήσεις που ακόμα συνδέονται με την παρακολούθηση των οξυδίων του θείου και η συμπερίληψη τέτοιων ρήπων αυτή τη στιγμή αναμφίβολα ε, θα καθυστερούσε και θα περιέπλεκε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παρακολούθηση και άλλων ρήπων δεν είναι πολύ σημαντική. Και θα θέλαμε την ενσωμάτωση στην προσέγγισή μας και άλλων ρήπων, όταν όμως αυτό καταστεί δυνατόν. Σε ό,τι αφορά το MRV, ε, Ω συμβολή στην Γενική Συμφωνία διατηρούμε τη θέση μα ότι πραγματικά η παγκόσμια αυτή η πρόοδος μέσω του IMO ε, θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό άξονα των προσπαθειών μας και θα πρέπει να επενδύσουμε και εμεί αυτή τη δικασία ούτως ώστε να συμπληρώσουμε ε, και να συμβάλλουμε περαιτέρω στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το σφαιρικό αυτό και παγκόσμιο αυτό καθεστώς. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την πρόταση που έχει ως στόχο να ευθυγραμμιστεί με τις ε, συζητήσεις που εξελίσσονται, όπου συνδέονται και συμμετέχουν η ΙΠΑ, Καναδά, η Ιαπωνία και ούτω καθεξής, για να ε, συζητήσουν το θέμα ε, αυτού του δικτύου επιχειρησιακής αποδοτικότητας. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ε, πάντα προτείναμε να συμπεριλάβουμε τα δεδομένα αποδοτικότητας στο πεδίο εφαρμογή ε, της πρότασής μας, γιατί εάν περιοριστούμε μόνο στο επίπεδο παρακολούθησης ε, στην παρακολούθηση των επιπέδων μάλλον του διευθυντήτου του άνθρακα, θα υπονόμευε τι περαιτέρω εξελίξει στι συζητήσει των IMO, όπου ακόμα επικεντρωνόμαστε στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια ανά σκάφος ε, και τη δημοσιοποίηση των δεδομένων MRV. Για μας ε, η διαδικασία αυτή παρακολούθησης υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης ε, θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα ως μέτρο πολιτικής. Εάν δεν δίνουμε πρόσβαση, εάν δεν ενημερώνουμε και τους επιχειρήσεις και τους καταναλωτές αλλά και το δημόσιο τομέα για αυτά τα δεδομένα, έτσι αφαιρούμε ένα από τα βασικά κίνητρα της πολιτικής μας. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για την ε, δράση, ούτως ώστε να κάνουμε τις πιο εύκολες και αποδοτικές επενδύσεις που ε, υπάρχουν στον τομέα και μπορούν να γίνουν στον τομέα μας. Ό,τι φορά τον περιορισμό σε δύο μεθόδους παρακολούθησης, έχουμε περάσει από τη λογική της ελαχιστοποίησης ε, των των διοικητικών διαδικασιών. Έτσι δεν υπάρχει νέο κόστος, νέος εξοπλισμός. Βασιζόμαστε στις εφιστάμενες πρακτικές ε, ανείχνευσης. Βασικό σημείο είναι επίσης το όριο. Εάν θα πάμε για τα 5.000 ή 400. Και εδώ τελικά πρόκειται για πολιτική απόφαση και επιλογή. Εμείς ε, θέσαμε τα επιχειρήματά μας για το όριο των 5.000, αρκετές ε, περιπτώσεις και θεωρούμε ότι οι 5.000 τόνοι είναι μία επιλογή που μπορεί να γίνει και σε διεθνές επίπεδο πάντα λαμβάνοντας υπόψη και το διοικητικό άχθος. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής δεν θεωρούμε ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα να γίνει πιο βραχή. Γιατί θα πρέπει ε, να υπάρξουν και πράξεις. πράξη. Ε, υπάρχουν αρκετές τεχνικές διατάξεις που θα πρέπει να διευθετηθούν ε, στο MRV. Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση σε αυτό το σημείο. Τέλος. Πολύ σύντομα για την αλλαγή της διαδικασίας ε, στη συνέχεια ως ένα διαφορετικό καθεστώς. Όταν ε, πήραμε το λόγο για πρώτη φορά, είπαμε ότι η χρήση εκτελεστικών και κατεξοδότηση πράξεων που προτείνονται στα MRV θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες διατάξεις της συνθήκης της αφώνας. Και κατεξοδότηση πράξεις προβλέπονται για ε, Τομεί όπου πρέπει να συμπληρώσουμε, να τροποποιήσουμε μη ουσιαστικά τμήματα τη πρότασης. Και πολλοί θεωρούν ότι η ελλαγή από το MRV να πάμε σε ένα καθεστώς κοστολόγησης, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ουσιώδες σημείο. Θα μείνω εδώ. Σας ευχαριστώ. Thank you, Michael. Ευχαριστώ, Michael. Ευχαριστώ καταρχήν για τη συνεργασία και για τις παρεμβάσεις σας. Σε κάποιες από αυτές σύντομα θέλω να απαντήσω, να τοποθετηθώ. Καταρχήν η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν ψήφισε ακόμα. Αλλά σκιαγραφούνται οι θέσεις που προηγούμενα περιέγραψα εγώ από πλευράς της. Ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετριόφρονα αλλά ρεαλιστική. Αυτό αναφέρεται πάντα. Αν είχαμε τέτοια πολιτική και στην αυτοκινητοβιομηχανία και τα εφαρμόζαμε, αυτά τα οποία είναι ρεαλιστικά, τότε θα είχαμε διπλάσιες σήμερα εκπομπές ρήπων. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τι γίνεται και χρειάζεται κάποιο θάρρος για να προχωρήσουμε. Και υπενθυμίζω ότι έχουμε αυστηρές τιμές σε σχέση για παράδειγμα με τον διάβλο, τη διόρυγα Βαλτικής ε, Βόρειας Θάλασσας και να δούμε και σε σχέση και τι θα γίνει και με για τη Μεσόγειο. Θέλουμε να υπάρχει θεμητό πλαίσιο ανταγωνισμού, ένα ισοδίκαιο πλαίσιο νομικό για όλους, να μην παραβιάζονται οι αρχές και σε σχέση με προσφυγές στο 10 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άλλες αποφάσεις ίσως θα μπορούσαν να ληφθούν. Θέλουμε δίκαιο ανταγωνισμό λοιπόν. Για το πεδίο εφαρμογής μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Τι θα ενταχθεί στο τέλος τέλος αν καταλήξουμε σε μεγάλο συμβιβασμό αν λέτε για παράδειγμα 4.900 ημέν και οι άλλοι 400 δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού αλλά σε σχέση με το 410 για παράδειγμα ίσως θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Έχετε δίκιο για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με την αλλαγή των κλιματικών προϋποθέσεων. Για την υγεία όμως δεν αληθεύει αυτό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα οξύδια του αζότου δεν διαδραματίζουν ρόλο και οι ασθένειες αυτές δεν είναι μεγάλης ε, σημασίας, μεγάλης εμβέλειας. Είναι σπουδαία τα στοιχεία αυτά, αυτά τα σημεία και πρέπει να δούμε με μείωση τι θα γίνει. Ωραίο είναι το επιχείρημα 98% το διοξίδιο του άνθρακα σε σχέση με όλα τα άλλα αέρια, αλλά και το 2% των υπόλοιπων αερίων κάνει και αυτό ζημιά. Ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξη και για το χρονοδιάγραμμα είμαι ανοιχτός και πρόθυμος να το κάνουμε πιο στενό, πιο σύντομο και για τροπολογία που ε, έχει κατατεθεί αν θα υπήρχε πλειοψηφία θα χαιρόμουν. Τώρα να, συμπεριληφθεί το, να συμπεριληφθούν τα οξύδια του αζότου θετικό και οι στόχοι μείωσης και αυτό σημαντικό και για την υποστήριξη θα ήταν λοιπόν σημαντικό να πετύχουμε αυτή τη μείωση και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάικλ. Να θυμίσω ότι αύριο θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και ε, στις 30 Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τώρα έχουμε την ε, έκθεση για την οποία είναι εισηγητής ο κύριος Λιμπεράτσκι, ρυθμίσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Φλίγκενστάιν θα πάρει το λόγο. Ναι, θα μιλήσω πολωνικά, μη φοβάστε, μια χαρά θα τα πω. Πρώτα απ' όλα, Εξ ονόματος του κυρίου Λιμπεράτσκι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις για την εξαιρετική, εξω, εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι θα στηριχτούν από την Επιτροπή οι συμβιβασμοί. Έχουμε 259 τροπολογίες, ε, ε, επί των οποίων έχουμε 19 συμβιβασμούς. Το ήδη από το 1990 ε, είχε γίνει δεκτή οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια, αλλά δυστυχώς από τότε δεν έχει τροποποιήσει. Συχνά οι καταναλωτές δεν ξέρουν τι είδους προστασία ε, μπορεί να έχουν σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Επομένως, είναι προφανές ότι η νομοθεσία πρέπει να επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να καλύπτονται και οι είδη ταξιδιού τα οποία δεν υπήρχαν ε, τον εποχή που εγκρίθηκε η οδηγία. Ο εισηγητής ε, της ε, Τράν έχει δύο στόχους Πρώτα απ' όλα η νέα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το όφελος των καταναλωτών από το υψηλό ε, ε, επίπεδο ε, προστασίας θα αυξήσει την ασφάλεια των αγορών και δεύτερον ότι θα υπάρχουν ίδιες συνθήκες για όλους όσους εμπλέκονται στην αγορά των οργανωμένων ταξιδιών και επίσης ότι ότι θα συμμορφούνται όλες οι ε, εταιρείε με τους στόχους αυτούς. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, προτείνει ο εισηγητής να διατηρηθεί το πλαίσιο της Επιτροπής με κάποιες προσαρμογές. Ε, καλεί λοιπόν ο εισηγητής να ληφθεί υπόψη και το κλικ όσον αφορά ε, τα οργανωμένα ταξίδια και επίσης ε, να υπάρξουν κάποιες προσαρμογές όσον αφορά τις ρυθμίσεις Link Travels. Όσον αφορά τώρα την εναρμόνιση οι σκιώδεις ηγητές συμφώνησαν σε στοχευμένη προσέγγιση εναρμόνισης που θα δίνει χώρο σε κάποιο βαθμό επικουρικότητα στα κράτη-μέλη. Κατά κάποιο τρόπο μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι το πεδίο αυτής της οδηγίας που προτείνεται εδώ δεν είναι αρκετά ευρύ. Ωστόσο, από το 1990 και ένθεν ο τουρισμός και η τουριστική αγορά έχουν αλλάξει. Οι προτιμήσεις επίσης έχουν ε, αλλάξει και επομένως νέα στοιχεία έχουν μπει στην αγορά. Ας πούμε ανεξάρτητα συμβόλαια για ενιαία ταξίδια δεν συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία. Οι οργανώσεις των καταναλωτών έχουν αναφερθεί σε πολλές ε, περιπτώσεις όπου ε, οι ε, καταναλωτές έχουν αγοράσει ταξίδι όχι από τον οργανωτή αλλά από κάποιον ενδιάμεσο και εκεί συχνά υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν ο εισηγητής προτείνει αυτού του είδους ε, ε, οι πωλήσει μεμονωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών είτε γίνονται από μεσάζοντα είτε από τον οργανωτή να διέπονται από το ίδιο καθεστώς. Μια ένα άλλο ε, πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να ότι έχουν πλέον αυξηθεί οι πωλήσει σε τέτοιων οργανωμένων ταξιδιών ε, από ε, ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία όμως αφορούν στην ουσία οργανωμένα μεμονωμένα ταξίδια θα πρέπει κατά την άποψη του ε, εισηγητού και προς ε, το συμφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών να ε, γίνουν σεβαστές οι συμβαστικές τροπολογίες. Αυτά είχα να πω εξ ονόματος του συναδέλφου Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, εξαιρετικά τα ισπανικά, τα ε, πολωνικά σας. Μας εντυπωσιάσατε. Ο κύριος Ριγάντας από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν κατανόησα, δεν κατάλαβα τα πολωνικά, αλλά κατάλαβα από πλευράς της ε, γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε και πρόεδρε δυστυχώ: είναι σημαντικό αυτό και νομίζω για όλους. Και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και να πούμε ότι για μια χώρα σαν την δική μου που έχει κύρια βιομηχανία τον τουρισμό έχει, είναι ένα κεφάλαιο ιδιαίτερης ε, σημασίας και προσοχής και οι ταχύς ρυθμοί με τους οποίους ε, εργαζόμαστε πριν από τις και σε σχέση με τους ε, συμβιβασμούς και συμβαστικές τροπολογίες πρέπει να δοθεί υποστήριξη στους όρους ε, προσέγγισης του κυρίου ε, Αυτό το οποίο θα ήθελα να πιστεύω είναι ότι θα είναι ακόμα δυνατόν ε, να μπορέσει να πάρει σάρκα και ωστά αυτή η φιλοδοξία και να καταλήξουμε σε, στο ότι έχει νόημα και έχει σημασία και είναι σωστό να γίνει αυτό. Στο τέλος πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στη δουλειά μας και πρέπει να προσπαθούμε να επιτύχουμε στόχους μέσα σε εύλογα χρονικά διαστήματα και γι' αυτό πρέπει τις υποχρεώσεις που έχουμε να τις επομισθούμε και να τις υλοποιήσουμε. Τώρα, σε σχέση με τον διάλογο που θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί, θα ήθελα εν πάση περιπτώσει να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπεράσχη για την προσέγγιση στα πολλαπλά και πολυσχηδή θέματα τα οποία τέθησαν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αληθεύει ότι αυτή η οδηγία είχε ξεπεραστεί και μπορούσε, έπρεπε να αντικατασταθεί. Οι νέοι, νέες συνήθειες των καταναλωτών, οι νέες χρήσεις μεταφορών, οι νέες ε, ε, πρακτικές καθιστούσαν παλαιά και ανεδαφική πλέον αυτή την οδηγία και θα έπρεπε λοιπόν να ανανεωθεί, να επικαιροποιηθεί σε σχέση με τις νέες πρακτικές και να εγγυάται κυρίως τα δικαιώματα των καταναλωτών τα οποία θα πρέπει να τα δούμε σε ένα ευρύτερο, πιο σύγχρονο πλαίσιο, αλλά και με πολλές εγγυήσει ε, νομικές ε, για τα δικαιώματά τους και να μην αφήνεται σε ένα εθελοντικό πλαίσιο σε σχέση με όσους εμπλέκονται. Και τούτων λεχθέντων προηγούμενα θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι ανεξάρτητα από την ταχύτητα εργασίας καταλήξαμε σε συμβιβασμούς. Συμβιβασμούς που νομίζω ότι είναι θετικοί και σε σχέση με την δυνατότητα διεύρυνσης αν μπορεί να γίνει είμαστε με ανοιχτό πνεύμα μπορούμε να δούμε προτάσεις συμβαστικές του εισηγητή και μπορούμε να τις συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να, κατα... να εγγυόμεθα μια υψηλότερο επίπεδο προστασίας των ε, ε, καταναλωτών και σε σχέση και με τις αγορές στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ε, εμπόριο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσει να γίνει αυτό. Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με τα παλαιά πρότυπα και υπάρχουν νέες πρακτικές, ε, νέες συνήθειες και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να προσαρμοστούμε σε αυτά. Και για το ε, σημαντικό θέμα των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων και σε σχέση και με τις προτάσεις δεν θα υπησέλθω σε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Ήθελα μόνο να σκιαγραφίσω κάποια πράγματα. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της ε, οδηγίας και το επίπεδο εναρμονισμού που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη το να μπορούν να υιοθετούν και αυστηρότερες διατάξεις. Ε, οι ορισμοί σε σχέση με τι ε, τις τουριστικές δραστηριότητες και για τις υπηρεσίες μέσα σε ένα λιγότερο αυστηρό πλαίσιο και μέσα στις ευθύνες που από το πλαίσιο αυτό απορρέουν. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό λοιπόν να τον και να ε, προαχθεί η αλληλεγγύη μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο δεν είναι δυνατό να αγνοούμε το, να υπάρχει δηλαδή η δέσμευση κάποιου συμβατική υποχρέωση και μετά να αγνοεί αυτή την υποχρέωσή του και το πώς θα μπορούσε να δράσει και ο καταναλωτής ε, όταν ε, ε, πρόκειται για τα δικαιώματά του θα πρέπει να μπορέσει να ζητήσει να είναι σεβαστά και να λαμβάνονται υπόψη. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε κύριε Σίγητα θεωρούμε χωρίς αμφιβολία ότι υπό τους όρους διατύπωσης των συμβιβασμών και αν είναι, θέλει ο εισηγητής να λάβει υπόψη και άλλα επιχειρήματα με χαρά να το δούμε. Τροποποιούνται λοιπόν με νέες ε, προτάσεις ε, για το διαδίκτυο και καλύπτονται ε, κενά τα οποία υπήρχαν νομικά. Και με ικανοποίηση μπορούμε να δούμε και να πούμε ότι δεν θα έλεγα να διαμαρτυρηθούμε, αλλά να εκφράσουμε όμως την θλίψη μας για την ταχύτητα και τη βιασύνη. Και σε σχέση και με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και την ιδιότητά μου ως σκιώδους εισηγητού, θα πρέπει να δούμε ότι ε, αυτή η ταχεία διαδικασία ε, πραγματικά πρέπει να μας κάνει να πούμε ότι θα πρέπει να ε, έχουμε αρκετό χρόνο να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να εξετάσουμε όλες τις πτυχές και να μπορέσουμε με καλές προθέσεις να είμαστε αποτελεσματικοί και με μια θετική πρόταση που ίσως ε, παραμένει εκτός ε, πλαισίου λόγω της ε, βιασύνης, λόγω της ταχύτητας ξέρουμε ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε και να εγκρίνουμε. Συμφωνούμε λοιπόν με το τμήμα εκείνο το οποίο είναι ουσιώδες, το ουσιωδέστερο πλαίσιο, ώστε να είναι βιώσιμος ο συμβιβασμός. Αν είναι όμως δυνατόν θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα ακούγοντας τις προτάσεις ε, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάισνερ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχήν τον εισηγητή τα οποία μας εξέθεσε από πλευράς του ο κύριος Φλέκενστάιν. Συμφωνώ και σε μεγάλο βαθμό με αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος Λιμπεράσκη και να δούμε ακριβώς το πεδίο εφαρμογής ε, επακριβώς. Και όταν αφορά, όσον αφορά τους κανονισμούς ε, click rules στο διαδίκτυο, σε μια, σε δέσμη μέτρων πρέπει να τα δούμε αυτά, αλλά να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτή τη σφαιρική αντιμετώπιση. Η μεταφορά για παράδειγμα δεδομένων ε, ονομάτων, στοιχείων από τη μία πλευρά στην άλλη ε, τότε λοιπόν αυτό θα πρέπει να μας κάνει να το θεωρούμε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενός πακέτου μέτρων, μιας δέσμης μέτρων. Όσον αφορά τις άλλες ρυθμίσεις ε, νομίζω ότι είναι κάπως ε, γενικόλογες. Αν μόνο ένα link ε, υπάρχει σε σχέση με μια εταιρεία εναέριων μεταφορών και όσον αφορά την μίσθωση οχημάτων θα πρέπει να δούμε κατά πόσον επαρκεί αυτό από πλευράς υπεύθυνου τρόπου κάλυψης των υποχρεώσεων. Αναφέρθηκαν λοιπόν τα στοιχεία αυτά τι σημαίνει ε, ο όρος υπηρεσίες. Ε, ε, σημαίνει διανυκτέρευση μαζί με το εισιτήριο των, της αεροπορικής εταιρείας. Υπάρχουν και κάποιες ε, ε, υπηρεσίες που εξαιρούνται από αυτήν την οδηγία, αλλά νομίζω ότι δεν ε, ανήκει αυτό μέσα στο πλαίσιο αυτό της συνολικής παροχής υπηρεσιών και έτσι θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Τώρα σε σχέση με το στοχευμένο, στοχοθετημένο εναρμονισμό θα πρέπει να είναι ένα πιο φιλο, καταναλωτικό πλαίσιο σε σχέση με, την, με τις προτάσεις. Δεν θέλουμε να παρακολύσουμε να είναι αποτελεσματικότερες για τους καταναλωτές οι ρυθμίσεις και από πλευρά των κρατών μελών πρέπει να υπάρξει και η προσαρμογή αυτή. Και πρέπει να δούμε για τις αυξήσεις τιμών αν με βάση την συμβατική υποχρέωση μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ξεπερνάνε ένα όριο 5% γιατί διαφορετικά κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια τέτοια κράτηση δεν θα μπορεί ίσως να χρηματοδοτήσει ε, τέτοιου είδους ε, ποσά, να τα καλύψει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Λίχτενμπεργκ, Εύα, σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτό ότι είναι απόλυτα αναγκαίο και κατεπήγον να καταλήξουμε σε μια επικαιροποίηση, ένα εξυγχρονισμό αυτού του πλαισίου, διότι υπήρξαν τεράστιες αλλαγές στη συμπεριφορά και τη στάση των καταναλωτών. Οι άνθρωποι σήμερα με τις κρατήσεις στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο ευέλικτοι από ό,τι στο παρελθόν. Βρίσκουν και συνθέτουν με ε, στοιχεία από διαφορετικές προτάσεις εκείνων που θέλουν να επιλέξουν. Και αυτό ε, οδηγεί και την και μια αλλαγή ε, στις ε, ευθύνες ε, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια λυσίδα ευθυνών. Πρέπει έτσι με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να υπάρξει σωστή αντίδραση και ο εισηγητής στους συμβιβασμούς του τα ουσιοδέτερα στοιχεία τα έχει συμπεριλάβει και μπορούμε να τα εγκρίνουμε και να τα δεχτούμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προσαρμοστούμε στους νέους τρόπους κράτησης ηλεκτρονικά. Υπάρχει η δυνατότητα τέτοιων προσφορών είτε μέσω ξενοδοχείων είτε ε, μέσω ταξιδίων που μπορούν ηλεκτρονικά να ε, γίνονται οι κρατήσεις με links, με διασύνδεση διανυκτερεύσεων ή και με ταξίδια τα οποία ε, ακολουθούν. Όλα αυτά θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο στην προστασία των καταναλωτών διότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πλαίσιο, το, η, μεγαλύτερη θα έλεγα αριθμητικά από πλευράς κρατήσεων πτυχή, η μεγαλύτερη συνιστόσα. Και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύεται ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν κάποιες αποσαφηνήσεις, επειδή κάποιες περιπτώσεις στην προστασία των καταναλωτών ε, δημιουργούν προβλήματα ή τριβές που πρέπει να αποσαφινιστούν επειδή ίσως οι ορισμοί δεν είναι απόλυτα σωστοί ή ακριβείς και γι' αυτό είναι αναγκαίο και σημαντικό οι ορισμοί να προσαρμοστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα λοιπόν, κυρίως όταν αφορά κάποιες αυξήσεις τιμών ή και κάποια μείωση από πλευράς ε, ποιότητας ή Κανείς δεν θα παραπονεθεί αν υπάρξει upgrading ξενοδοχείου στην προσφορά των ταξιδιωτών, γιατί η αναβάθμιση η ποιοτική είναι καλό. Είναι όμως πρόβλημα αν κάποιος έχει κρατήσει, έχει κάνει κράτηση για ένα ταξίδι και προβλέπεται διανυκτέρευση σε ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων ή κάποιων αστέρων και καταλήγουμε στο να ε, υπάρχει πρόβλημα με το λουτρό στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει σημαντικές αποσαφηνήσεις να γίνουν Ιδιαίτερα σημαντικό είναι με βάση τα βιώματα και την πείρα που συλλέγουμε από πλευράς δημοσιευμάτων είναι να βρούμε σωστές ρυθμίσεις σε περίπτωση πτώχευσης, σε περίπτωση ε, που κλείνουν κάποιες επιχειρήσεις. Να βρεθούν δυνατότητες ε, οι όσοι έχουν κάνει κρατήσεις ε, να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, να μπορούν να ταξιδέψουν και να μπορέσουν να καλύψουν το ταξίδι τους αυτό. Είναι σημαντικό να βρεθούν τέτοιες ε, λύσεις σε συνδυασμούς ε, και να δούμε και στις ανταποκρίσεις και συνδυασμούς να υπάρξουν σωστοί ορισμοί, ώστε οι καταναλωτές να προστατεύονται και να μπορούν να αντιδράσουν έγκαιρα για να προστατευτούν τα, συμφέροντά τους. Αποφασιστική σημασία είναι να ενημερώνονται και να πληροφορούνται για τις αλλαγές ε, οι καταναλωτές όταν γίνονται αλλαγές και τότε και το ίδιο το επίπεδο προστασίας ε, αλλοιώνεται και πρέπει να υπάρξει κάποια αντίδραση. Τώρα όλα αυτά είναι εφικτά και μπορούν να γίνουν ώστε οι καταναλωτές, γυναίκες και άντρες να μπορούν να διασφαλίζουν τα αναγκαία επίπεδα προστασίας ε, των συμφερόντων τους. Εδώ νομίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μπορούσαμε σε μεγαλύτερο βάθος να, εξετάζαμε αυτό το θέμα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο, τον Λίσαντα, που είπε ότι ταχαίως εργαστήκαμε. Έπρεπε όμως να υποβληθεί μια πρόταση και να υπάρξει μια ρύθμιση γιατί διαφορετικά θα υπήρχε καθυστέρηση. Υπάρχουν ήδη σημαντικές αλλαγές και προστίθεται και κάποιο άλλο θέμα το οποίο όπως και ο συνάδελφος έτσι και όταν προέρχεται κάποιος από μια περιοχή που έχει τουριστική ένταση και ε, έχουμε και επιχειρήσεις ε, που στην χώρα προέλευσης ε, παρέχονται και όταν έχουμε αρνητικές προσφορές κάποιες προσφορές που δεν τηρούν τα υπεσχημένα ή απαραμελούμε την προστασία των καταναλωτών, ε τότε δημιουργούνται στο τέλος προβλήματα και πρέπει στην χώρα προορισμού να επιλύονται τα προβλήματα. Εκεί δημιουργούνται προβλήματα για τους ταξιδιώτες και όχι στη χώρα προέλευσής τους. Αυτό είναι λοιπόν ένα πρόβλημα για τις χώρες στόχους να δούμε τις ρυθμίσεις αν αυτές δεν ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημένα τι θα πρέπει να γίνει και πώς να αντιδράσουμε. Πρώτον, στα ταξιδιωτικά πρακτορία και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να αποσαφινιστεί ότι πρέπει ο αθέμητος ανταγωνισμός να αποκλειστεί και να μπορούν να τηρούνται τα υπεσχημένα και να μην παραμένουν, ας το πω έτσι, εγκαταλειμμένοι κάποιοι ταξιδιώτες στη χώρα προορισμού τους. Αν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ένας τουρίστας, ας το πούμε έτσι, ε, εγκαταλείπεται από το γραφείο ταξιδίων ή την επιχείρηση που τον έχει στείλει εκεί, πρέπει κάτι να γίνει. Υπενθυμίζω δηλαδή τις χώρες εκείνες που έχουν μεγάλη τουριστική δραστηριότητα και όπου ο τουρισμός έχει μεγάλο ρόλο. Πρέπει να μεριμνήσουμε το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών να είναι υψηλό, αναβαθμισμένο, ώστε κατά τις διακοπές τους οι ταξιδιώτες αυτοί να μπορούν να προστατεύονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τις διακοπές τους και την αναβαθμισμένη ποιότητα που έχουν για τους ανθρώπους. Εκταμιεύουν οι ε, πολίτες, ε, ε, μαζεύουν χρήματα για να περάσουν τις διακοπές τους όπως επιθυμούν και πρέπει να μπορούν να προστατεύονται ώστε να ανταποκρίνεται η προσφορά με την αρχική προσφορά στο επίπεδο που έχει περιγραφεί και το οποίο εκείνοι έχουν κλείσει, έχουν κάνει κράτηση. Είναι σημαντικό, είμαστε Επιτροπή Τουρισμού και πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Είμαι όμως ικανοποιη... ικανοποιημένοι με τις συμβαστικές προτάσεις και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Thanks, Chairman, and thanks to the... Η κυρία Τζάκη Φώστερ, ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή και τον συνάδελφο που έκανε την παρουσίαση. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε η αρμόδια επιτροπή, άρα δεν αποφασίζουμε μόνοι μας. Ωστόσο, γνωμοδοτούμε και γενικώ ε, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε αυτήν την επικαιροποίηση. Να σας πω ότι έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα από, μία από τις πιο, πιο μεγάλες αγορές ε, ταξιδιών και ε, επομένως ε, υπάρχουν ένα σωρό νέες applications οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα των ταξιδιών. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες όσον αφορά τους ορισμούς και επίσης όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Επιπροσθέτως, αυτή η διασύνη, και δεν επικρίνω εδώ τον εισηγητή. Ε, είχαμε κανονίσει κάποιες συναντήσεις ε, οι οποίες ε, όμως συγκλήθηκαν τελευταία στιγμή και οι περισσότεροι βουλευτές δεν μπορούσαν να παραστούν. Οι σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων ή οι ε, βοηθοί μας έπρεπε να είναι ε, παρόντες γιατί εμείς δεν μπορούσαμε αλλά δεν μπορούμε να ασκούμε τέτοια πίεση πάνω στους ε, συνεργάτες μας θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε συναντήσεις όπου μαζί με τους άλλους συναδέλφους από τις άλλες ομάδες να κάνουμε μια πραγματική διαπραγμάτευση η Κομισιόν έκανε μια πρόταση, δεν απήντησε στις ερωτήσεις τις οποίες ε, ε, είχα υποβάλει σε αυτήν ε, κατά τη διάρκεια της ακροάσεως της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Είχα αναφερθεί σε κάποιες περιπλοκότητες οι οποίες παρουσιάζονται την στιγμή της κράτησης online. Βεβαίω, εμεί θέλουμε να βρούμε ένα σωστό τρόπο αναθεώρηση όλων των πεπαλαιωμένων στοιχείων. Επίσης ε, ε, πρέπει να πω ότι όσον αφορά, uh, ε, όσον αφορά και το standalone έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και η Κομισιόν δεν έχει διάθεση και ούτε φαίνεται να την ενδιαφέρει πάρα πολύ όσον αφορά το κλίμα και επίσης και εδώ έχουμε ένα ε, ζήτημα το οποίο ε, μας απασχολεί. Ε, λοιπόν, ε, προσπαθεί ας πούμε ένας πελάτης, ένας αξιδιώτης να κάνει κράτηση σε μια αεροπορική εταιρεία και ξαφνικά βγαίνει με ένα κλικ ένας σύνδεσμος που τον πηγαίνει σε ε, κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο και μετά ένα, ένα άλλο ε, πρωτόκολλο μπορεί να το ξαναφέρει στην ε, αεροπορική εταιρεία στην οποία ήθελε να κλείσει αρχικά εισιτήριο. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα μπλέξιμο όσον αφορά τα θέματα αυτά. Και η επικουρικότητα παίζει ρόλο εδώ. Νομίζω ότι κάποιοι από τους συναδέλφους ήδη αναφέρθηκαν στα κάποια από τα προβλήματα εδώ. Ε, σίγουρα είναι πάρα πολύ βεβαρημένο το πινακιό μας με το απόγευμα. Δεν έχουμε και πάρα πολύ αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η διαδικασία είναι ικανοποιητική. Είναι κρίμα, είναι κρίμα ε, γιατί περνάμε πράγματα ε, τα οποία δεν έχουν αποσαφινιστεί. Μας πιέζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν προχωρήσει όπως έχει το κείμενο αυτό, τελικά οι καταναλωτές θα την πληρώσουν. Θα είναι οι ασθενείς κρίκοι για μία ακόμα φορά. Εδώ δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για το 261 ή κάτι παρόμοιο. Δεν είμαστε ερασιτέχνες. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το πράγμα και αυτή είναι η κατι παρομοιο δεν ειμαστε ερασιτεχνες νομιζω οτι ολοι γνωριζουμε πω λειτουργει το πραγμα και αυτη ειναι η θεση μα. Δεν θέλω να πω κάτι επικριτικά για τον ε, εισηγητή. Προσπαθεί και αυτό να κάνει ό,τι μπορεί. Ξέρουμε ότι ε, έχει καταλήξει σε συμβιβασμού, αλλά ωστόσο δεν πιστεύουμε ότι έχουν ε, λυθεί όλα τα προβλήματα και ούτε πιστεύουμε ότι οι πληροφορίε είναι σαφεί και ούτε πιστεύουμε ότι και η Κομισιόν έχει ίδια τη τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα τα οποία είχαμε υποβάλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να πω μόνο ότι εμείς ε, δεν είμαστε η κύρια ε, καθήλυν αρμόδια επιτροπή. Ακολουθούμε μόνο ένα χρονοδιάγραμμα που μας έχει επιβάλει η Επιτροπή ΙΜΚΟ. Όμως ε, για να είμαστε και δίκαιοι προς αυτούς είναι άλλη ακόμα, μία ακόμα ε, περίπτωση όπου η Επιτροπή καθυστερημένα υπέβαλε νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο. Εμείς εδώ καιρό τη ζητούσαμε την πρόταση. Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Ξέρουμε ότι και στη δική μας ε, Επιτροπή τα πράγματα πάνε έτσι, καθυστερούν και αυτό μετά δημιουργεί προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα ο εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη, μπορεί να μα εξηγήσει γιατί υπάρχουν αυτέ οι καθυστερήσει από πλευρά Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίω ε, δεν μπορώ να σχολιάσω επί των διαφόρων ε, συμβιβασμών επειδή δεν του έχω δει. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα βεβαίω ε, θα γνωρίζετε ότι είναι περίπλοκο το θέμα με πολλές διαφορετικές απόψεις που εξέφεραν ε, διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Και είχαμε μακροσκελείς, εκτενέστατες διαδικασίες διαβούλευσης και δική μας πρόθεση ήταν ε, να έχουμε μια ισορροπημένη πρόταση κατόπιν αυτών των ε, παρεμβάσεων που ακούσαμε κατά τη διάρκεια του γύρου διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη στήριξη που άκουσα από πολλούς ε, συναδέλφους ε, για το έργο της Επιτροπής που νομίζω ότι είναι μια εφικτή και ισορροπημένη πρόταση λαμβάνοντας υπόψη και τις διεστάμενες απόψεις που είχαμε. Είχαμε τους ε, καταναλωτές από τη μία, τη βιομηχανία από την άλλη και όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους. Αυτό εξηγεί σε έναν βαθμό και το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, δεν μπορώ να σχολιάσω επί των συμβαστικών προτάσεων, όμως από πλευράς της Επιτροπής να σας πω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και, τους, ε, και τον διπλό στόχο της ε, πρότασης. Αφενός θέλουμε να επιτύχουμε υψηλό επίπεδο προστασία ε, του καταναλωτή σε αυτό το τομέα και από την άλλη έχουμε και την άρση των εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο που βεβαίως ε, απαιτεί ένα αλφα επίπεδο εναρμόνισης. Ιδάλλως ε, και οι εμπορευόμενοι, οι οικονομικοί φορείς θα έχουν δυσκολίες κατά την ε, άσκηση της δραστηριότητά τους όταν ας πούμε υπάρχει διαφορετική διαφορετικές απαιτήσει και υποχρεώσεις ό,τι αφορά την πληροφορία. Αυτό του δημιουργεί πρόβλημα στην ε, διασυνοριακή, στο διασυνοριακό εμπόριο. Ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ο κύριος Φλέκενστάιν, ο κύριο Λιμπεράσκη, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θα διαβιβάσω στον κύριο Λιμπεράσκη τα σχόλια και τι παρατηρήσει σα. Κύριε Ντεγκράντες, εμείς είμαστε που το επιτρέπουμε να γίνεται αυτό με μας. Δηλαδή με τέτοια ένταση χρονικά και τέτοια πίεση να συζητούμε και να εξετάζουμε τέτοιες προτάσεις. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι στο μέλλον δεν θα πρέπει να το δεχόμαστε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε αύριο, όπως ξέρετε, και μετά στην ΕΜΚΟ η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου και νομίζω ότι ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί για την Ολομέλεια, αλλά νομίζω πάει 14 Μαρτίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Έχει το λόγο ο κύριος Γκρός. Μάλιστα, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εδώ πάλι πιέζει ο χρόνος με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πρώτα όλους τους συναδέλφους <clears throat> και που τις κοινοβουλευτικές ομάδες και οι εισηγητές για την πραγματικά επικοδομητική συνεργασία. Δεν είναι βέβαια κάποια ιδανική λύση. Έχουμε διαφορετικές προτάσεις ενώπιον μας και μια πρόταση που σύντομα θα ήθελα να επεξηγήσω η πρόταση αυτή βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεταξύ εκείνου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στην Επιτροπή Ένβη, Επιτροπή Περιβάλλοντος και αυτά που άλλοι συνάδελφοι στην Επιτροπή προτείνουν και έχει ως εξή το θέμα. Η Επιτροπή προτείνει, έχει υποβάλει αυτή την πρόταση <clears throat> να ακολουθήσουμε την πρόταση Stop the Clock ώστε μετά από το 2014 να βρούμε το πεδίο εφαρμογής ε, μεταγενέστερα. Αυτό που οδηγεί. Οδηγεί στο ότι η δική σας κοινοβουλευτική επιτροπή βρίσκεται στα δύο ακραία. Η μεν να σταματήσουμε σε σχέση με το 2020, η άλλοι να υπάρξει ε, η ένταξη προτάσεων στο διεθνές επίπεδο ενώ άλλοι συνάδελφοι έλεγαν ότι πρέπει να υπάρξει μια ε, δυνατότητα ε, δράσης Τώρα για να σας πληροφορήσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ότι θα είχαμε το σύστημα μέχρι το 2014, μετά θα είχαμε μέχρι το 2016 μια επιθεώρηση, ανα, επανεξέταση και μετά υστερότερα θα είχαμε το τελικό ε, σύστημα το οποίο θα ίσχυε. Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και φυσικά η πρόταση που έχουμε μπροστά μας και που δεν ε, ε, υποστηρίζεται πρέπει να υπάρχει μια πρόταση συμβιβαστική που θα διασφαλίζει ένα ασφαλές πλαίσιο αλλά και την ελαστικότητα που είναι αναγκαίο να υπάρχει. Και σε σχέση με την δική μας προσέγγιση υποβάλλεται μια πρόταση που με το σύστημα Stop the Clock θα διασφαλιστεί μέχρι το 2016 και με τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν συλλαγεί σε παγκόσμιο επίπεδο είτε θα τηρηθεί αυτή η πορεία είτε όχι ανάλογα με τις προτάσεις που θα έχουν ε, ε, υποβληθεί ώστε να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο δράσης. Τα προτερήματα τα πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης θα ήταν το είτε θα είχαμε μια σαφή ευρωπαϊκή λύση, αλλά ακόμα καλύτερο μια σαφή διεθνή ρύθμιση που θα ήταν ακόμα καλύτερη ως ε, εναλλακτική δυνατότητα για να μπορούσαμε σε σχέση με το 2016 να κάναμε κάτι τελευταίο τώρα ε, για τις περιφέρειες ε, στις εσχατιές ε, έχουν υποβάλει διάφορες προτάσεις συνάδελφοι. Προσπαθήσαμε το συμβιβασμό να τον λάβουμε ως εξή υπόψη ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω άλλες εναλλακτικές λύσεις και από πλευράς του συνόλου της ε, διαδρομής να υπάρξει μια, ένας τρόπος υπολογισμού ώστε να μην είμαστε ε, μη συνεκτικοί. Προτείνουμε λοιπόν ε, και για τη δεύτερη φάση εδώ στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο να λάβουμε την πρώτη φάση που θα εφαρμοστεί υπόψη και στις διεθνείς πτήσεις ε, ούτως ή άλλως ε, δεν θα λαμβάνονται αυτές, ε, αυτές οι διεθνείς πτήσεις υπόψη μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή είναι η συμβαστική πρόταση λοιπόν. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω ότι στο ένα ή άλλο σημείο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν αποτελεσματικό συμβιβασμό για να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα, ιδιαίτερα όσον αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Χαντράουι. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για το έργο του και για τη συμβαστική πρόταση που έχουμε επιτάπητος. Ε, Βεβαίω είναι ένα φάκελο που έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και ξέρουμε ότι και οι συνάδελφοί μας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουν μια πιο ριζοσπαστική θέση. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχει φιλοδοξία μέχρι την επόμενη ε, συνεδρίαση του ΙΚΑΟ να καταλήξουμε σε παγκόσμια συμφωνία. Ε, που θα εφαρμοστεί μέχρι το 2020. Και νομίζω ότι αυτές ε, οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να πάνε στον να καλύτερα, να δώσουμε όσο να το περισσότερες ευκαιρίες, γιατί είναι και ο στόχος μας. Ε, θέλουμε η πολιτική αεροπορία και η αεροναυτιλία να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι χρήσιμο ότι αυτό το stop the clock που έχει ήδη ξεκινήσει να το συνεχίσουμε ως προσέγγιση μέχρι να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε και μια πίεση να φροντίσουμε το ώστε και όσοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ε, να γνωρίζουν ότι εμείς θέλουμε πραγματικά να υπάρξει συμφωνία Γι' αυτό η πρόταση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσουμε με αυτή την προσέγγιση του εναέριου χώρου, δηλαδή όλες οι πτήσεις που περνούν ε, από τον ε, Ευρωπαϊκό εναέριο Χώρο να λαμβάνονται υπόψη. Και αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα. Να διατηρήσουμε λοιπόν ε, πίεση. Να λάβουμε υπόψη για κάποιες εξαιρέσεις που έπρεπε να έχουμε για κάποιες ευρωπαϊκές ε, επικράτειες. Είναι λογική αυτή η συμβαστική πρόταση και ταυτόχρονα διατηρούμε και κάποιες αρχές ε, που έχουμε συμφωνήσει. Ως ομάδα θα ε, στηρίξουμε την πρόταση, εκτός από τους συναδέλφους που ίσως είναι πιο κοντά στους πρασίνους, όμως νομίζω ότι συνολικά θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστούμε τον συναδέλφο Γρόσου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάιστερ. vielen Dank auch. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ματιέ Γκρός γιατί επελήφθη αυτού του σημαντικού θέματος ε, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Οι χώρες που συνέρχονται σε συνόδους για την προστασία του κλίματος και λαμβάνουν ε, ε, τέτοιες καλές αποφάσεις κρίμα το ότι από πλευράς ΑΙΚΑΟ, από πλευράς ΔΟΠΑ, Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει μια, ένα χρονοπλαίσιο στο οποίο προτάθηκε. Μέχρι το 2016 θέλουν να εκπονηθεί μια τέτοια πρόταση. Δεν είμαστε βέβαιοι αν αυτό θα λειτουργήσει έτσι, αλλά θα αναμένουμε και θα προσδοκούμε ότι θα υπάρξει μια τέτοια πρόταση. Και όταν υπάρξει μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιδρώσουμε. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση του Μάτιο Γκρός. Διότι δεν πρέπει να υπονομευθούν τα πράγματα, να βιαστούμε από πλευράς Ευρώπης με κάτι το οποίο δεν θα υποστηριχθεί ε, σε παγκόσμιο πλαίσιο και θα αγνοηθεί και πρέπει να υπάρξει ευκαιρία στη διεθνή κοινότητα να εξευρεθεί μια λύση και ταυτόχρονα και θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα και να δείξουμε ότι αν δεν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα εμείς θέλουμε να δοθεί συνέχεια σε αυτό το εγχείρημα ώστε αυτό το πρότυπο να είναι μια καλή εναλλακτική δυνατότητα ώστε να ασκηθεί πίεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει το stop the clock να σταματήσει το χρονόμετρο, να σταματήσει όχι μέχρι το 2016 αλλά μέχρι το 2020. Αλλά συνολικά αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος Γκρός νομίζω είναι ένας καλός συμβιβασμός και μπορούμε να τον δεχθούμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Κυρία Λίχτενμπεργκ, ευχαριστώ θερμά. Αυτό το συμβιβασμό με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να τον υποστηρίξω. Για ένα απλό λόγο. Την τελευταία φορά όταν συζητήσαμε το θέμα και ε, εγκρίναμε το, την πρόταση Stop the Clock να σταματήσει το χρονόμετρο, είπαμε αυτή θα είναι μια προθεσμία, μια διορία. Μετά δεν θα υπάρξει άλλη υπεραιτέρω επέκταση. Πρέπει να αντιδράσει η διεθνής κοινότητα μέχρι τότε. Εσείς επαναλαμβάνετε τώρα το ίδιο πράγμα αλλά με πρόταση παράτασης τι σημαίνει αυτό για τους εταίρους με τους οποίους διαπραγματευόμαστε. Να σταυρώσουν τα χέρια τους σημαίνει αυτό και να μην κάνουν τίποτα. Και η Ευρώπη θα παρατείνει βήμα προς βήμα με κλιμακούμενο τρόπο τις προθεσμίες. Έτσι στέλνουμε το λάθος μήνυμα όμως. Στέλνει το μήνυμα η Ευρώπη αν το δεχτεί αυτό ότι όταν υπάρχει κάποια αντίσταση στο διεθνές πλαίσιο ε, τότε υπακούμε προσαρμοζόμαστε και προχωρούμε. Λάθος είναι αυτό λοιπόν. Έχουμε λάβει μια απόφαση, ήδη στην διαμόρφωση λήψης απόφασης ε, είχε αποδυναμωθεί, διότι πολύ καλύτερο θα ήταν να είχαμε ένα πρότυπο λύσης ε, όπου με ένα συνεκτικό πλαίσιο θα συνδεόντουσαν όλα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, άλλη ιστορία. Νομίζω κάτι κάνουμε στραβά εδώ ή εσείς κάνετε κάτι στραβά, διότι όλους αφαιρείται κίνητρα από όλους που θα μπορούσαν να ήταν σύμμαχοί μας στην παγκόσμια κονίστα, στην παγκόσμια σκηνή και υπάρχουν άνθρωποι που λένε πρέπει να κάνουμε κάτι για να μειωθούν ε, οι εκπομπές ρήπων στις εναέριες μεταφορές. Όπως και στον τομέα των οδικών μεταφορών και στη βιομηχανία και στο επίπεδο ρήπων γενικότερα. Αυτοί οι εταίροι και ε, σύμμαχοι τώρα απογοητεύονται από αυτή τη στάση μας. Όταν ακούν ότι η Ευρώπη όταν υπάρχει κάποια αντίθεση ή αντίσταση παρατείνει τις προθεσμίες ούτως ή άλλως απογοητεύονται και είμαι πεισμένη ότι αν προτείνετε αυτό έτσι εσείς τώρα και την άλλη φορά θα ακουστεί πάλι «Α, δεν αντέδρασε η διεθνής κοινότητα, εμείς θα προσαρμοστούμε πάλι και θα δώσουμε νέα παράταση». Λάθος αυτό, λάθος. Είναι αναγκαίο να είμαστε συνεπείς και σταθεροί στις θέσεις μας. Και σε σχέση με την ε, προθεσμία της Επιτροπής Περιβάλλοντος να επεκτείνουμε τα χρονικά όρια θα ήταν λάθος. Δεν πρέπει να γίνει δεν πρέπει μόνο τα συμφέροντα των επιχειρήσεων να λαμβάνουμε υπόψη, αλλά σφαιρικά όλα τα στοιχεία. Τι τι προκαλεί και δημιουργεί η αλλαγή η κλιματική και ποιες είναι οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν ότι αν τώρα είπα η Κίνα, η Ινδία, οι άλλοι στη Νότια Αμερική δεν ανταποκρίνονται και δεν εγκρίνονται άμεσα, δεν εγκρίνουν άμεσα, αυτό το ξέραμε και πιο πριν ότι δεν θα το ενέκριναν αμέσως. Και δεν συμφωνώ λοιπόν να του στείλουμε το μήνυμα ότι όταν υπάρχει κάποια αντίθεση ή αντίσταση, ε, τότε η αντισταση τοτε σκύβει το κεφάλι, γονατίζει και δίνει παράταση προθεσμίας. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τους ε, φορείς μεταφορών και climate change, αλλαγές δηλαδή κλιματικές σε σχέση με τις ε, μεταφορές μας. Πρέπει να δράσουμε και να δράσουμε αποτελεσματικά, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, μην λαμβάνουμε μόνο βραχυπρόθεσμα στοιχεία υπόψη σε σχέση με τις μεταφορές. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον Μάθιου Κρός. Ήταν δύσκολο το έργο του για να βγει κάποιο νόημα σε αυτήν την υπόθεση. Να ξεκινήσω από αυτό. Γιατί πολλά τμήματα ε, των συμβαστικών τροπολογιών αποτέλεσαν αντικείμενο τη ε, επικοδομητική συνεδρία που είχαμε την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη εβδομάδα μπορούμε να τη στηρίξουμε. Όμω η δυσκολία είναι ότι το όλο ζήτημα είναι μια συμβαστική τροπολογία. Υπάρχουν λοιπόν τμήματα που έχουμε διαφορές. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μία ε, μονομερή προσέγγιση. Εκεί καταλήγουμε τελικά. Και ουσιαστικά άμα μεταφέρουμε τώρα την προθεσμία και μετά πάλι δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Το ίδιο κάνουμε. Εμείς έχουμε προβάλει δύο τροπολογίες, μία εγώ προσωπικά, που ουσιαστικά λένε ότι ελλείψη ε, πραγματικής αντικτύπου για το προτινόμενο πρότυπο του ενέργειου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ε, αδυναμία ε, συμφωνίας ε, στην ε, ολομέλεια της Διεθνής Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, που ε, απαιτεί κάποιες υποχρεώσεις από αυτές τις χώρες πριν εφαρμοστεί το σύστημα, αν υποβληθούν τέτοια μέτρα σε τρίτες χώρες και η έλλειψη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις πτήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή ε, αυτής της οδηγίας θα πρέπει να ανασταλεί επαόριστον. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Αποδεχόμεθα ότι ε, συνεχίζεται αυτή η προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του Stop the Clock και νομίζουμε ότι υπάρχει εδώ θέμα. Γιατί είναι ενάντια στον ανταγωνισμό. Έχουμε και εμείς μικρές ε, αεροπορικές εταιρείες που τις ε, μπλέκουμε σε όλη αυτή την υπόθεση και θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα τουλάχιστον μέχρι το 2016. Δεν το ζήτησαν οι ίδιες εταιρείε αυτές και ο κανονισμό ποτέ δεν έλεγε ότι μιλούσαμε για το ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Η Επιτροπή μιλούσε για το σύνολο. Και αυτό μας θέτει σε δύσκολη, δυσχερή θέση, γιατί τελικά θα κάνουμε αυτό το stop the clock και θα επανέλθουμε στον αρχικό κανονισμό. Αυτό είναι προφανές. Και οτιδήποτε για να αποφασίσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι δικό της θέμα. Όμως ε, ένα στοιχείο ακόμα για την μετάβαση στο, στο μοντέλο του ενέργου χώρου. Δεν είχαμε αξιολόγηση αντικτύπου. Εγώ έχω μιλήσει με πολλά ενδιαφέρομενα μέρη και η μετάβαση από τον αρχικό κανονισμό στις πτήσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το μοντέλο του ενέργειου χώρου. Λοιπόν, από όλου ε, με όσου συνομίλησα, κανένα δεν θεώρησε από τον χώρο τη βιομηχανία ότι πρόκειται για καλή ιδέα. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το κόστο, αν θα είναι πιο ε, επικερδές ή ε, κοστοβόρο για τι εταιρείε και για του ε, επιβάτε. Δεν τα έχουμε λύσει λοιπόν και απαντήσει αυτά τα ερωτήματα γιατί η Επιτροπή είναι απελπισμένη, θέλει μεταμανίας να ε, έχει αποτελέσματα, γι' αυτό και θέλει να μας μπλέξει και εμάς όλη αυτή τη διαδικασία για το Κοινοβούλιο. Επομένως, στηρίζουμε πολλά από τα όσα μας προτείνει ο Μάθιου. Ουσιαστικά θέλουμε όλα να σταματήσουν και μετά το 2016 να επανέλθει ο ΙΚΑΟ. Εμείς δεν έχουμε με παγκόσμια συμφωνία εάν πράγματι αυτοί θεωρούν την καλύτερη επιλογή. Όμως αυτή τη στιγμή, Πρόεδρε, βρισκόμαστε μεταξύ σκύλες και χάρευδης και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Μάθιου, δεν ξέρω αν μπορούμε να εξετάσουμε αυτή τη συμβαστική πρόταση, να αφαιρέσουμε κάποια τμήματα γιατί με πολλά συμφωνούμε. Εκεί που λέτε για την αξιολόγηση δεκτύπου είναι μόνο για ένα παράρτημα. Εμεί θέλουμε κάτι παραπάνω από ένα παράρτημα για να θίξουμε το ζήτημα τη αξιολόγηση ε, δεκτύπου στον εναέριο χώρο και πώ ε, θα το μετρήσουμε. Θέλουμε να μπει στο διατακτικό με πολύ ισχυρότερη θέση για να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Αυτά είχα να πω από πλευράς της ομάδας μου, Πρόεδρε. Και πάλι να ευχαριστήσω τον Μάθιο που πραγματικά κατέβαλε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να καταλήξει σε κάποια αποτελέσματα εδώ και περιμένω ε, με αδειμονία τα αποτελέσματα. Εσείς μην περιμένετε πάντως Ευχαριστώ πρόεδρε. Ουσιαστικά θα ήθελα μια πιο διαφανή, μια λιγότερο γραφειοκρατική διεθνή λύση με βάση τις προτάσεις της ΑΙΚΑΟ του ΔΟΠΑ θα έπρεπε να έχουμε το stop the clock μέχρι το 2020. Λογικό θα ακούγονταν αυτό. Η δουλειά όμως που έκανε ο Ματιο Γκρός είναι πολύ καλή και γι' αυτό θα υποστηρίξω το συμβιβασμό που μας προτείνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας πω ότι δεν είναι δεν συνηθίζεται να χωρίζουμε σε τμήματα τις ε, τροπολογίες ε, συμβιβασμού. Ε, αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Μπάντρομ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου τα οποία σχολίασαν επί του θέματος. Ιδιαίτερος δε ε, ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Γκρόσο για την ε, προσπάθειά του να έχει επικοδομητική προσέγγιση και προσπάθεια να επιλύσει τις διαφορές. Η Κομισιόν παραμένει σταθερή στη θέση της. Θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές αντικατοπτρίζει την θέση έτσι όπως ακούστηκε στην ε, συνέλευση της ΣΑΙΚΑΟ αλλά και επί σειρά ετών ε, από τα χείλη των εκπροσώπων των μεγάλων αεροπορικών ε, επιχειρήσεων. Δηλαδή όλοι οι εμπλεκόμενοι στον φορέα θέλουν αυτήν την προσέγγιση αυτοί που λένε ότι τεχνικώς κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, πολλές φορές έχουμε κάνει τα δύνατα δυνατά και ξέρουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ περιορισμένο ε, διοικητικό κόστος ή ε, επιπλοκή. Γιατί βεβαίως ε, ξέρουμε ότι ε, και η Eurocontrol έχει ε, πολύ προχωρημένα εργαλεία όσον αφορά, την, ε, ε, τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων. Έχουν γίνει πολλές αξιολογήσεις αντικτύπου όσον αφορά αυτήν την ε, προσέγγιση και από την ΑΕΚΑΟ αλλά και εμείς έχουμε κάνει ε, με εκτενή αξιολόγηση της ε, προσέγγισης εναερίου χώρου. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλη αξιολόγηση αντικτύπου εάν θεωρείτε ότι είναι απολύτως απαραίτητη. Διατηρούμε τη θέση ότι η πρότασή μας και τεχνικά και νομικά στέκει. Ωστόσο, εκτιμούμε και τις απόψεις ε, οι οποίες ε, θεωρούν ότι θα πρέπει ε, να μελετηθούν και περαιτέρω δυνατότητες διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος παρανόησης. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η επιλογή πεδίου προσφέρει, παρέχει προστιθέμενη αξία. χωρίς να αποκλείουμε θετικά στοιχεία και στην προσέγγιση ε, εκτός του εναερίου χώρου. Βεβαίως είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιες ε, ρήτρε αναθεώρησης υπάρχουν, ποια είναι η διασύνδεση της δικής μας νομοθεσίας ε, με τις διατάξεις της ΑΙΚΑΟ. Αυτό είναι αντικείμενο πολιτικής συζήτησης και εν πάση περιπτώσει αυτό που αποτέλεσε την ε, τελική μας ε, θέση ήταν ε, να χαμηλώσουμε λίγο τις περιβαλλοντικές μας απαιτήσεις περιμένοντας σε αυτή την ενδιάμεση δηλαδή περίοδο την επίτευξη μιας διαδικασίας πιο ολοκληρωμένης και σας διαβεβαιώ ότι το 2016 θα έχουμε την αξιολόγηση του αποτελέσματος που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε με την πλήρη ευθυγράμμιση. δεν είδαμε τα συμβαστικά κείμενα, γι' αυτό δεν μπορούμε να σχολιάσουμε λεπτομερία, αλλά πραγματικά θα θέλαμε ε, να διαβάσουμε τα κείμενα αυτά, να έχουμε στενή συνεργασία με όλους ε, τους εμπλεκόμενους ε, και τους συμμετέχοντες σε την διαβούλευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ο κύριος Γκρός, μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Και όλες οι παρεμβάσεις κατέδειξαν ότι αυτά που πάνε υπερβολικά μακριά για τους μεν δεν πάνε αρκετά μακριά για τους δε. Και ένα συμβιβασμός πρέπει να πει κανείς ότι πρέπει να τον δει ως συμβιβασμό. Δεν μπορεί όλοι να ικανοποιηθούν απόλυτα. Και έχουμε και στον συμβιβασμό και την αρχή του earmarking, του προκαθορισμού της χρήσης κονδυλίων και αυτό πρέπει να, αναπτυχθεί στο, στο πιο αποτελεσματικό πλαίσιο. Δεν είναι θέμα μόνο του να εισπράττονται κάποια χρήματα, αλλά για τη σωστή τους χρήση. Και κάποιες παρατηρήσεις τώρα σε σχέση με ε, τον, την προλαλή σας, κυρία Φώστερ. Κάνει λόγο για μελέτες επιπτώσεων, impact assessment. Δεν είναι μόνο αυτό εδώ, Τζάκι, αλλά και στο άρθρο 28, εδάφιο 7, που σαφώς λέγεται ότι οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από μια εξειδικευμένη μελέτη επιπτώσεων. Λοιπόν, η μελέτη επιπτώσεων Ευχαριστώ. Πρέπει να το δούμε λοιπόν το ότι εντάσσεται σε σχέση με το ίδιο το άρθρο. Ήταν σαφώς ε, ε, η δική μας επιθυμία αυτή και ελπίζουμε ότι αύριο θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν ήταν μόνο εσωτερικά εδώ συμβιβασμοί δική μας αλλά και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αξίζει λοιπόν έτσι να δούμε σε σχέση με την πρόταση αυτή μια λύση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι βιώσιμη. Ευχαριστώ λοιπόν όλους. Πρόεδρος, αύριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και η Επιτροπή ΕΝΒΗ θα ψηφίσει την 30 Ιανουαρίου. Επόμενο θέμα είναι το ΣΕΣΠΛΙΣ 2. Οι συγητές ε, είναι απόντες. Οι συντονιστές μήπως είναι εδώ. Φαίνεται ο κύριος Μπρογκρός θα μιλήσει ε, εξ του κυρίου Μαρινέσκου μόλις τελειώσει τη συζήτηση που έχει για το ETS με την κυρία Φώστερ, τον βλέπω ότι έχει ξανακαθίσει και γι' αυτό τώρα μπορεί να μας πει ποια είναι η άποψη του κυρίου Μαρινέσκου για το θέμα. Σε συνδύο. Κύριε Γκρός. Πολύ γρήγορα πήγαν πρόεδρε αυτά. Εντάξει, λοιπόν. Δεν θα τα διαβάσω ρουμανικά, εντάξει. Ο συνάδελφος Μαρινέσκου προσπάθησε να τα μεταφράσει και λέει το πιο σημαντικό σε σχέση με τις τροπολογίες είναι η υποστήριξη της ρύθμισης σε σχέση με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και σε σχέση με τις τροπολογίες και με την ε, ανεξαρτησία των ε, εθνικών αρχών σε σχέση με την ε, πιστοποίηση θα πρέπει να επιτευχθεί συμβασμός λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση που υφίσταται στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει η υποστήριξη να υπάρχει μία αρχή που θα έχει κοινέ ευθύνε σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Υποστηρίζει λοιπόν σε σχέση με αυτή τη γνωμοδότηση ότι θα πρέπει να εδράζεται σε μια απόφαση και για το ε, προτιμόμενο αυτό, ε, την προτιμόμενη προσέγγιση προτείνεται να διοργανωθεί με ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστή, με ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, ώστε να υπάρξει η αναγκαία συμφωνία, να υπάρχει μια εταιρική σχέση. Θα έλεγα αμέσω μετά από όλα αυτά και έτσι κερδίζουμε χρόνο σε σχέση με τη γνωμοδότηση λέγοντας ότι ως ΕΛΚ με την έκθεση αυτή θέλουμε να τηρήσουμε την πίεση ώστε να μπορέσει από πλευράς Ευρώπης ε, να προχωρήσει το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να ε, δοθεί εντύπωση ότι παρεκκλίνουμε από αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να το απαιτούμε περαιτέρω. Έχουμε νομοθεσία όπου τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν δεν τα υλοποίησαν, δεν ήταν πρόθυμα να προσαρμοστούν. Το πιο σημαντικό λοιπόν ο στόχος είναι να σταλεί ένα μήνυμα από το Ευρωκοινοβούλιο ότι αυτό θέλουμε να επιτευχθεί Όλα τα άλλα για μια ε, ρυθμιστική αρχή, για μια ευρωπαϊκή αρχή είναι ένα περαιτέρω θέμα που μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό από πλευράς Μαρινέσκου για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι μια κοινή συζήτηση γιατί οι συγγετέ είναι οι ίδιοι, οι σκιώδεις. Επομένω, να δώσουμε το λόγο και για την έκθεση του κυρίου Σασόλη αλλά και για την έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου έχετε το λόγο. Α, εντάξει, περίπλοκα. Πρώτα στα γαλλικά για την έκθεση του Νταβίδ. Ο Νταβίδ δεν μπορεί να είναι εδώ για λόγους υγείας για την έκθεσή του. 85 τροπολογίες επιβλήθησαν, μεγάλο τμήμα αυτών ε, έγιναν δεκτές. Ε, μόνο μία συμβαστική τροπολογία υπάρχει για την διακυβέρνηση. Για τις ε, τροπολογίες που επευλήθησαν, 29, 30 και 31 του Ζάκη Φώστερ, για ε, τις Τζάκι Φώστερ ε, δεν είμαστε υπέρ. Δηλαδή η αφαίρεση των στρατιωτικών αρχών είναι η παναχώρηση με κίνδυνο για την ασφάλεια. Τώρα, για 40, 41 και 42. Εκεί ο Νταβίτ θα ήθελε να υπαλληθεύσει με την Επιτροπή τι συμβαίνει, γιατί ε, έτσι με αυτές τις τροπολογίες αφαιρείται ο ορισμός κάποιων όρων ε, και του πεδίου εφαρμογή των κατεξοδότηση πράξεων. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν ε, πιο προσεκτικά. Η τροπολογία 12 του Νταβίτ έχει αποσυρθεί, δεν ισχύει πλέον. Και μετά υπάρχουν αρκετέ τροπολογίε του κ. Μαρινέσκου, οι οποίες επιβλήθησαν, που αφαιρούν την τροποποίηση του όρου κράτος μέλος και την αντικατάστασή του με τον όρο αρμόδιες αρχές. Για την διακυβέρνηση προτείνει ένα συμβασμό που λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής με την τροπολογία του Νταβί, της Τζάκη Φώστερ και του Σίμψον. Ε, διατηρούμε τον όρο Executive Board που συνάδει και με τον ε, τη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. Όμως θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι αυτές οι αρμοδιότητες ε, αφορούν κυρίως τη συνδρομή προς τον εκτελεστικό διευθυντή κατά την προπαρασκευή προετοιμασία αποφάσεων που θα ληφθούν στο Management Board, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το εκτελεστικό συμβούλιο μπορεί να ε, πάρει απόφαση μόνο όταν υπάρχει αναστολή ε, της ε, ιδιότητας του διευθυντή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με πλειοψηφία 5 από τα 7 μέλη τουλάχιστον. Βεβαίω ευρύνουμε τη σύνθεση με έναν πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, ε, πέντε μέλη αντί για τρία για μια ε, διετή θητεία με δυνατότητα αναθεώρησης, ανανέωσης. Αυτά για την έκθεση του Ντάβιντε. Τώρα πολύ σύντομα για την έκθεση Μαρινέσχου. Τρία σημαντικά σημεία. Πρώτον, συμφωνούμε ότι πρέπει να έχουμε πιο αυστηρά ε, συστήματα επιδόσεων με δυνατότητα κυρώσεων και ισχυρότερο ρόλο της Επιτροπής. Έτσι θα έχουμε λιγότερες καθυστερήσεις, μεγαλύτερη ασφάλεια, χαμηλότερο κόστος, αλλά και ο ανθρωποκεντρικός παράγοντας ε, επανισάγεται Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για μας. Δεύτερον, για τις ε, υποστηρικτικές υπηρεσίες, εδώ αυτό μας ανησυχεί γιατί υπάρχει ένας διαχωρισμός μια διαίρεση αυτών των υπηρεσιών και μας απασχολεί τι θα γίνει ε, στον, στην κοινωνική διάσταση. Και γι' αυτό έχουμε αφενός ε, αυτά τα σημεία και αφετέρου, πέραν αυτών των ανησυχιών, πρέπει να μας απασχολήσει και η ε, αποδοτικότητα. Και τέλος, για τις εθνικές εποπτικές αρχές, είναι σαφές ότι υπάρχουν προβλήματα με αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κάποιες φορές δεν υπάρχουν αρκετές κυρώσεις ή δεν, δεν έχουν το απαραίτητο δυναμικό. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα και να ενισχύσουμε τις εποπτικές αυτές αρχές. Αυτά σε αδρές γραμμές ε, οι παρατηρήσεις ε, του Σκιώδους ε, για την έκθεση Μαρινέσκου. Ευχαριστούμε κυρία Σα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μαρινέσκου. Στο Στρασβούργο είχαμε μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών όπου αρκετά πράγματα μπορέσαμε να συζητήσουμε. Τώρα, σε σχέση με τους συμβιβασμούς ε, που συμφωνούμε με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί πράγμα το οποίο είπε και ο κύριος Γκρόσο, ότι η δομή θα πρέπει να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Δεν θα πρέπει να διαλυθεί, να αποδιαρθωθεί αυτή η δομή. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε πού υπάρχουν συνεργασίες εκτός ΦΑΠΣ και που για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό μπορούν να, να προχωρήσουν το έργο και να μην ε, δημιουργηθούν προβλήματα. Υπάρχουν συνεργασίες που λειτουργούν καλά και μπορούν να διασφαλιστούν και πρέπει αυτό να διασφαλιστεί. Τώρα όσον αφορά την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών, καλό είναι να συμπεριλαμβάνεται αυτό το στοιχείο και μια και σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ έχω μια ερώτηση που, για την οποία δεν έχω κάποια απάντηση. Από την ομάδα μου τίθεται το ερώτημα τι γίνεται με το Γιβραλτάρ. Η νομική υπηρεσία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει να δούμε τι θα γίνει με το Γιβραλτάρ και πώς αντιμετωπίζεται. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Yeah, Με το Γιβραλτάρ είναι πάνω από τις δυνάμεις μου, κυρία. Μάλιστα, ευχαριστώ. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, για μένα πολύ σύντομα υπάρχουν δύο ουσιώδη στοιχεία. Το ένα, έχω την εντύπωση σε κάποιους τομείς όπως το unbundling ή ο διαχωρισμός ότι έχουμε ιδεολειπτική προσέγγιση, μια ιδεολογική προσέγγιση με πολύ λίγη, ας το πω έτσι, αναφορά στην πραγματική πραγματικότητα και στην πραγματική πρακτική. Πρέπει να βρεθεί μια σωστή αντικειμενική λύση. Το να βρούμε τεχνητές ε, διαχωριστικές γραμμές ε, δεν ε, οδηγεί πουθενά, δεν είναι επωφελές. Δεύτερο, πιστεύω ότι Στη συνολική αυτή σύνολη συζήτηση για τον ε, ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, Single European Sky, όχι μόνο θέματα ασφάλειας πρέπει να εντάσσονται, αλλά θέματα κλίματος ε, και ιδιαίτερα ε, θέματα περιβάλλοντος ιδιαίτερα με την εξοικονόμηση ανάλογα με τον φορέα μεταφορών ενέργειας και αυτό θα ήταν ένα σημαντικό στοιχείο θα έλεγα θα έπρεπε με σοβαρό τρόπο να αντιμετωπιστεί αυτό σοβαρό στοιχείο στη συνολική συζήτηση. Δεύτερο, στην τροπολογία 26 για το, την αιτιολογική σκέψη 2, την σύγκρουση συμφερόντων στην ίδια την ΕΑΣΑ, την αναφέρουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ένα πολύ σημαντικό σημείο θα έλεγα αυτό. Αυτό που θέλουμε είναι και εδώ αηφορία να διασφαλίζεται στην κλιματική πολιτική και στην περιβαλλοντική μας πολιτική με έναν ε, τρόπο που θα έχει εμβέλεια για το πρόβλημα των delegated acts, των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Έχουμε την τάση μέχρι κάποιες δηλώσεις όλα να ρυθμίζονται με, κατεξουσιοδότηση, ε, με, με πράξεις κατεξουσιοδότηση. Σε κάποιους τομείς όταν πρόκειται για καθαρά τεχνικά μέτρα αυτό ίσως δικαιολογείται. Όμως υπάρχει γενικότερα η τάση και πολιτικές αποφάσεις με κατεξουσιοδότηση πράξης ε, να καλύπτονται. Και στο τέλος τέλος το Κοινοβούλιο να μην έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην λήψη απόφασης αυθεντικά με, σε βάθος συζητήσει και αναλύσεις. Αφαιρείται η δυνατότητα αυτή από το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είμαι κατά της τάσης της πολλαπλής χρήσης ε, των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Και στις, ε, στους σκιώδεις εισηγητές αυτά έχουν ήδη συζητηθεί. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο λόγια όσον αφορά την έκθεση σας όλοι. Ναι, γιατί κάνουμε και τις δύο εκθέσεις μαζί, ναι. Σχετικά με την έκθεση σας όλοι, λοιπόν. Γενικώ θεωρούμε ότι οδηγείται προς τη σωστή κατεύθυνση ο εισηγητής στο μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης. Ωστόσο υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας προβληματίζουν. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρόταση αλλαγής ονόματος από ΕΑΣΑ σε EAA, ανώφελο, Επίσης, το ζήτημα σχετικά με το Executive Board. Δεν συμφωνούμε με οτιδήποτε ε, δεν προβλέπει συμμετοχή και δική μας ε, σε αυτό το board οποιοδήποτε κι αν είναι, οποιοδήποτε συμβούλιο δεν έχει δική μας εκπροσώπηση, ε, δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνος. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη βεβαίως. Βεβαίως αυτό είναι πρόταση που προέρχεται από την Επιτροπή. Επίσης, σχετικά το να γίνει η NSA, NAA, αυτό επανέρχεται και στην έκθεση Μαρινέσκου. Νομίζουμε ότι κάποιες ε, τροπολογίες οδηγούνται προς την εσφαλμένη κατεύθυνση και θεωρούμε ότι ε, αποτελούν βάρος για τη διαδικασία και θα ε, οδηγήσουν σε σύγχυση. Επίσης να πω ότι εμείς και ως ομάδα ε, πραγματικά ενστερνιζόμαστε αυτή την ιδέα του Ευρωπαϊκού Ανοιχτού ε, Ουρανού γιατί πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει να προωθηθεί το ζήτημα αυτό. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως και ο κύριος Σασόλη προσπαθεί ε, να ε, συγκεράσει πολλές απόψεις. Όσον αφορά την έκθεση Μαρινέσκου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ε, για την έκθεση. Κοιτάξτε αυτές οι εκθέσεις είναι τεχνικές, δεν είναι τόσο απλές και εύκολες αλλά και εδώ έχουμε ένα ζήτημα παρόμοιο όσον αφορά το NSA που θα γίνει NAA Έχω συζητήσει με τους εμπλεκόμενους φορείς στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ξέρετε, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτές οι δύο αρχές, δηλαδή αν μιλάμε για την αρχή του κράτους μέλους ή αν μιλάμε για την ενιαία ε, αρμόδια αρχή, δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επίσης, όσον αφορά το σχεδιασμό του εναερίου χώρου, ε, αυτός αναλαμβάνεται από τις ε, ANSPs. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι εδώ θα πρέπει να επιλεγεί η διαδικασία επιτροπής μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Όσον αφορά την εισαγωγή νέου οικονομικού ρυθμιστού, χωρίς πρώτερη συζήτηση και χωρίς να ξέρουμε τι είδους οικονομική regulation θα υπάρξει, δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνο. Επίση, Επίσης, οποιοδήποτε διαχωρισμός ε, δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνος γιατί δεν έχει γίνει πρώτερη διερεύνηση αγοράς. Τέλος, δεν θέλω να ε, δημιουργώ προβλήματα επί αμφιλεγωμένων ζητημάτων, αλλά ε, όσον αφορά το Γιβραλτάρ υπάρχουν πολλές τροπολογίες σχετικά με την ε, εφαρμογή του ανοιχτού ουρανού στο Γιβραλτάρ. Είναι προφανές ότι πρόκειται εδώ, το Γιβραλτάρ δηλαδή είναι βρετανικό έδαφος και επομένως δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα ε, που να μην λαμβάνει αυτή την κατάσταση ε, και να μην αναγνωρίζει την κατάσταση αυτή. Ε, υπάρχουν και τροπολογίες εδώ από συναδέλφους δεξιά μου που δεν καταλαβαίνω γιατί ενδιαφέρονται για το Γιβραλτάρ αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν υποβάλει τροπολογίες. Ε, δεν καταλαβαίνω ότι, ε, γιατί θα πρέπει να συζητιέται το θέμα αυτό και στην έκθεση Μαρινέσκου και στην έκθεση όλοι. Υπάρχει σχετική συμφωνία, έχει γίνει αποδεκτή από όλους. Ξέρω ότι γενικώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σε αυτές τις εκθέσεις και εμείς το ίδιο, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε πράγματα τα οποία είναι απαραδεκτά. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Όπω σα είπα και προηγουμένω, είναι περίπλοκε οι εκθέσει και γι' αυτό ευχαριστούμε του συναδέλφου Μαρινέσκου και σα όλοι. Έχω τους συντονιστές, ε, θα πρέπει, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρία των συντονιστών πιο γρήγορα, επομένως ε, δεν χρειάζεται να φύγετε, θα αρχίσουμε σε λίγο. Ο κύριος Δεγκράντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε προς εμάς, Πρόεδρε, δεν θα σας φανεί τόσο περίεργο όπως φαίνεται στην κυρία Φώστερ να ρωτάει κανείς για το Γιβραλτάρ. Και μάλιστα σε σχέση με την κυβέρνηση της Ισπανίας το ερώτημα τι συνέβαινε με το Γιβραλτάρ και τις διαφορετικές στάσεις που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ρυθμίσεις για τον εναέριο χώρο. Μόλις εγκρίναμε στην Επιτροπή μας τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικυρώθηκε αυτό σε σχέση με τη διακήρυξη του Λονδίνου ε, και δεν υπήρχε καμία αναφορά για, την, για θέματα κυριαρχίας, αλλά εγώ θα το αναφέρω. Οι διαφορές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας είναι παλαιές σε σχέση με την ε, συνθήκη της Ουτρέχτης και έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μας και δεν θέλουμε αυτές να τις θολώσουμε, να τις ε, κυλιδώσουμε, αλλά σε σχέση με αυτό το θέμα είναι πολύ απλός ο λόγος. Υπήρχε μια ρήτρα που επαναλαμβανόταν σύμφωνα με την ε, διακήρυξη του Λονδίνου που έλεγε ότι η εφαρμογή των ρυθμιστικών διατάξεων για τον εναέριο χώρο σε σχέση με το Γιβρατάρ ε, θα αρθούν μέχρι ότου υπάρξει συμφωνία μεταξύ των μερών Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια αξιολόγηση υπέρ του ενός ή του άλλου, αλλά απλώς αναφερόταν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα και έπρεπε να επιληθεί. Υπήρξε μετά η διακήρυξη, η περιβόητη διακήρυξη της, Κόρδοβα, της Κόρδοβας και όπως ε, υπήρξε η διακηρυξη η περιβοητη διακηρυξη της κορδοβας και οπως υπηρξε η απαντηση προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, ε, υπήρξε ε, μια ας το πω και πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στη διακήρυξη του Λονδίνου. Αυτή είναι η νομική κατάσταση του θέματος. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θέσει την διακήρυξη του Λονδίνου στα δικαιώματα επιβατών και την διακήρυξη του, της Κόρδοβας στο θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Γιατί αυτό είναι αντιφατικό αν γίνεται έτσι. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Για το θέμα της ε, κυριαρχίας τώρα εδώ δεν είναι ε, περί αυτού. Είναι το να επανέλθουμε στον ορθολογικό τρόπο αυτής της εφαρμογής ε, της ε, ε, αποκαλούμενης διακήρυξης του Λονδίνου που λέει ότι έρεται η εφαρμογή μέχρι ότου υπάρξει συμφωνία που θα καταλήξουν τα δύο μέρη. Συνεχίζονται λοιπόν αυτές οι, δια, και σε σχέση με αυτή την δήλωση δεν είναι μεροληπτική και πρέπει λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι να επιληθεί το θέμα με μια ε, σολομόντια λύση ε, αλλά να δούμε το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με το 140. 146 148 σε σχέση με τη δήλωση διακήρυξη του Λονδίνου που έχει νομικά πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εφαρμογής και λέμε ότι έρεται η εφαρμογή αυτών μέχρι ότου οι δύο χώρες θα προβούν σε διάλογο ώστε να μπορέσει να ρυθμιστεί το θέμα αυτό το οποίο αφορά το, το αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Baldwin τώρα. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους ε, βουλευτές ε, που μίλησαν σαφώς και έκαναν κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Και εγώ μια παρατήρηση ε, να κάνω. Ας δούμε τι ακριβώς είναι το ΣΕΣ συν 2, αυτή η δέσμη. Είναι μια συγκεκριμένη, περιορισμένη δέσμη προστίκη στην ήδη υπάρχουσα δεν πρόκειται για μια ε, μεγάλη και συνολική ε, αλλαγή της πολιτικής, ούτε και μια νέα ιδεολογική τοποθέτηση απέναντι στις διατάξεις. Κυρία Λίχτεμπερ, και το είπατε αυτό, πρέπει να πω ότι συμφωνώ τόσο με αυτά που είπατε ε, για το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι λαμβάνουμε αρκετά υπόψη την σοβαρή διάσταση και τη σοβαρή παράμετρο του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλές ε, και διαφορετικές τροπολογίες. Προσπάθησα ε, να τις ομαδοποιήσω όσον αφορά την, ε, τις τροπολογίες επί της εκθέσεως σας όλοι όσον αφορά την ΕΑΣΑ πρώτα και μετά ε, τις τροπολογίες επί της εκθέσεως του κυρίου Μαρινέσκου, Μαρινέσκου για τον ενιαίο ουρανό. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες διαγράφουν ε, το, από, τον, από το πεδίο εφαρμογής ε, τα στρατιωτικά αεροδρόμια. Πρέπει να πω ότι έχουμε την αίσθηση ότι η πρόταση βασίζεται τελικά σε μία ε, παρεξήγηση. Αυτό που προσπαθούμε είναι να ευθυγραμμίσουμε την ΕΑΣΑ με αυτά που βρίσκονται ήδη στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό του 2002. Υπάρχει ήδη ανάγκη και απέτηση πιστοποίησης ε, όταν έχουν και το εντός αγωγικών General Air Traffic επομένως ε, δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί. Ο κύριος Γκρός αναφέρθηκε στην έννοια του φόβου κατακερματισμού των αρχών των κρατών μελών. Ε, η ιδέα ήταν ε, αντιθέτως να συνδυάσουμε τις αρμόδιες αρχές ε, των, σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αντιτιθέμεθα καθόλου η την αλλαγή της ορολογίας στην οδηγία σε ΕΑΣΑ. E Όμως θα, θεω, θα προτιμούσαμε την έννοια competent authority, αρμόδια αρχή. Γιατί κάθε χώρα ξέρει ποια είναι η αρμόδια αρχή. Μερικές φορές είναι όντως οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, μερικές φορές όμως είναι κάποιος άλλος φορέας. Γι' αυτό προτιμούμε τη δική μας προσέγγιση, τη δική μας διατύπωση, αλλά συμφωνώντας μαζί σας ότι θα πρέπει να αποφευθεί οποιοδήποτε, κατακερ... Ε, οποιοδήποτε κατακαιρματισμός. Όσον αφορά ε, ο, τον φορέα πιστοποίησης των εθνικών αρχών, αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά πιστεύουμε ότι εδώ πραγματικά χρειάζεται σοβαρότατη ε, μελέτη αντικτύπου. Θα θέλαμε να επανέλθουμε αργότερα στο θέμα αυτό, γιατί αυτή η πρόταση είναι λίγο πρόημη σε τούτη τη φάση. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ήθελα να θίξω όσον αφορά το θέμα της ΕΑΣΑ. Περνάω τώρα στο θέμα του ΣΕΣ. Είχαμε πολλές τροπολογίες, πολλές φορές εκ διαμέτρου αντίθετες. Όσον αφορά το ζήτημα των ορισμών, των υφιστάμενων ορισμών. και των σχετικών ζητημάτων, είναι γεγονός ότι οι προτινόμενες ορολογίες της τροπολογίας 149, 151 και 153 ευθυγραμμίζουν κάποιες, ε, ε, ε, ευθυγραμμίζουν κάποιες ορολογίες και επομένως μπορώ να τις καλωσορίσω, αλλά μπορώ να σας εξηγήσω γιατί το 2004 κάναμε κάποιες ε, ε, αλλαγές. Οι ορισμοί την προηγούμενη δεκαετία χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν ευρύτατα ε, και αν τώρα ξανακάνουμε αλλαγές τότε θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα χωρίς να αποκλείονται και κάποιες νομικές επιπλοκές τις οποίες τώρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Επίσης, μετά την τροπολογία 160 και μετά έχουμε πολλές τροπολογίες όσον αφορά την αρμόδια αρχή. Ε, πρέπει να πω ότι είναι γεγονός ότι ταυτίζουμε ε, σε αυτό το επίπεδο την ε, οδηγία με την ασφάλεια και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην περιμένουμε πρώτα να γίνουν ατυχήματα και μετά να αντιδράσουμε το ζήτημα των support services, των υπηρεσιών υποστήριξης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έδειξε τουλάχιστον ένας ομιλητής. Πρέπει να αναφέρομαι εδώ ε, στην τροπολογία 2.14 αλλά ε, και με τις τροπολογίες μέχρι τη 2.56. Είναι γεγονός ότι ενδεχομένως ε, η πρότασή μας λίγο πιο φιλόδοξη και επίσης ε, εμείς αρχικά προτείναμε ε, να διαχωριστούν οι υπηρεσίες πυρήνα από τις υπόλοιπες ε, υπηρεσίες αλλά στην ουσία είναι δύσκολο για τους νέους εισαγόμενους στην αγορά να παρέχουν υπηρεσίες σαν main provider τούτου λεχθέντος συμφωνούμε απολύτως ε, ότι συμφωνούμε με την εισαγωγή στο συμβαστικό κείμενο της έκφρασης με την προϋπόθεση ότι θα επιλεγεί η πιο συμφέρουσα ε, πρόταση του main service provider. Επίσης από τη 2.37 μέχρι τη 2.79 προσπαθήσαμε ε, να απαντήσουμε με πιο συγκεκριμένα ε, κείμενα ε, και δεν είμαι σίγουρος ότι οι τροπολογίες προσφέρουν κάτι παραπάνω. Τα προτινόμενα μέτρα ε, σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν ήδη, δεν έχουν, αυτό μπορώ να το δεχτώ, δεν έχουν δώσει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε τη δεύτερη περίοδο αναφοράς να την αφήσουμε στους έξι μήνες και ωστόσο μπορούμε να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι όσον αφορά ε, το πρόγραμμα γενικά. Επίσης αναφέρθηκε ο ανθρώπινος παράγων. Η τροπολογία 320 αναφέρεται στη δημιουργία συμβουλευτικής ομάδας. Συμφωνούμε με αυτά που λέτε όσον αφορά τη σημασία του πράγματος αλλά για λόγους ε, διοικητικής ε, ε, αποτελεσματικότητας θα θέλαμε να αφήσουμε τον, αυτόν τον ανθρώπινο παράγοντα στην, στις ομάδες διαβούλευσης και στην κοινωνική διαβούλευση που προβλέπεται ήδη. Αυτά είναι κάποια στοιχεία πρώτα Μπορούμε βεβαίως να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε γενικές γραμμές ε, δεχόμαστε τις τροπολογίες. Το θέμα του Γιβραλτάρ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι απλώς μπορώ να ε, σημειώσω προσεκτικά το θέμα αυτό ε, και συγγνώμη που μιλάω και αγγλικά λέγοντας κάτι τέτοιο θα λάβω υπόψη μου και αυτά που είπε η κυρία Φώστερ και αυτά που είπε ο κύριος Κανάλης. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά διάλειμμα λέει ο Πρόεδρος μέχρι να ξεκινήσει στις πέντε ακριβώς η συνεδρίαση των συντονιστών. Ε, μία μικρή διακοπή λοιπόν έτσι ώστε να φύγουν όσοι δεν είναι συντονιστές από την αίθουσα.